Συνάδελφοι, έχουμε πολύ γεμάτη μερίσια διάταξη με δύο πολύ σημαντικές ακροάσεις. Γι' αυτό είναι καλό να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας, αν και έχουμε αρχίσει να κουραζόμαστε. Είναι πολύ έντονες συζητήσεις, αλλά τα πλονεκτήματα, ε, το πλονέκτημα μάλλον το να έχουμε σε μια μισή μέρα τους εκπροσώπους όλων αυτών των αρχών ε, αρμόδιων για την έγκριση τύπου είναι πολύ θετικό. Υπάρχουν ε, βέβαια ταυτόχρονα πολλέ συνεδριάσει και ψηφοφορίε σε άλλε επιτροπέ. Γι' αυτό βλέπετε συναδέλφου να παίρνουν βγαίνουν στην αίθουσα. Πάντω είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί. Σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Λοράν Βερνό και την κυρία Μπεατρή Λοπέ, που είναι ε, διευθυντέ της, ε, του ομίλου Ταξεράμ της Γαλλίας. Θα σας δώσω το λόγο για να κάνετε κάποιες αγωγικές παρατηρήσεις. Ε, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είμαι Γενικός Διευθυντής της Ιούτα Κασεράμα. Πρόκειται για μια ιδιωτική ε, γαλλική εταιρεία, ανεξάρτητη, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις δοκιμές επιστοποίησης για τη, για τη Γαλλία και θα σας δείξω σε λίγες διαφάνειες ποια είναι η ομάδα μας ώστε να καταλάβετε καλύτερα τι ακριβώς κάνουμε. Ελπίζω πως όλοι θα βλέπετε τις διαφάνειες περίπου. Πρόκειται για περίπου 400 ε, μηχανικούς και τεχνικούς, 200 ε, δοκιμές ε, γύρω από το Παρίσι, Έχουμε το 20% του κύκλου εργασιών μας γίνεται με διεθνείς, σε διεθνείς εγκαταστάσεις, μία στην Κίνα και μία στην Ρωσία και ε, συνεργαζόμαστε με 40 περίπου χώρες. Έχουμε δύο μεγάλες εγκαταστάσεις γύρω κοντά στο Παρίσι. Ε, πρόκειται, ε, είμαστε οι πρωτοπόροι στις κατηγορίες πιστοποίηση 1 και 1. Τώρα, σύντομες ιστορικές, ε, ιστορικά στοιχεία. Ε, έχουμε ξεκινήσει το Λινάζ Μοντερί που είναι ένας ιστορικό, ένα ιστορικό μέρος όπου έχουν, ε, υπάρχει συγκεκριμένη πίστα και έχουν σπάσει πολλά παγκόσμια ρεκόρ αλλά εκεί έχουν γίνει και οι πρώτες εργασίες όσον αφορά την κατανάλωση αλλά και τα κουτιά ταχυτήτων που εκεί κάπως σταθεροποιήθηκαν. Η ΟΤΑΚ δημιουργήθηκε το 1945, η ε, εταιρεία για την οποία μιλάμε, και έχει εργαστήρια τα οποία είναι εγκατεστημένη στον χώρο του Λινάς Μοντλερή. Θα δείτε και κάποιες φωτογραφίες από εκεί και μετά ε, αγοράσαμε ε, το 2008 και τις εγκαταστάσεις στο Μόρφοντεν στο Βόρειο Παρίσι. Είμαστε Ασχολούμαστε κυρίως με ε, τα οχήματα που τρέχουν στους δρόμους. Ε, βέβαια πρόκειται για γεωταχή, αλλά όχι μόνο για τα γεωταχή. Συνεργαζόμαστε με Γάλλους κατασκευαστές κυρίως, αλλά όχι μόνο. Με Γερμανούς, με Άγγλους, Ιάπωνες, Κινέζους και άλλους. Ε, συνεργαζόμαστε με πολλούς κατασκευαστές εξοπλισμών και στο... εργαζόμαστε επίσης στον κόσμο των γεωργικών μηχανημάτων, των στρατητικών εξοπλισμών, λοιπόν ε, δουλεύουμε δηλαδή με ό,τι έχει να κάνει με οχήματα, με τροχούς στην Ευρώπη. Έχουμε διάφορες, διάφορους κλάδους. Ο βασικός είναι η ρύθμιση και η πιστοποίηση. Ε, και εδώ η κυρία Λοπές είναι υπεύθυνη για αυτό το τμήμα των κανονισμών και της πιστοποίησης και θα είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Επίσης έχουμε ένα μεγάλο τμήμα το οποίο ασχολείται με τις δοκιμές και την εμπειρογνωμοσύνη, δηλαδή είναι τα εργαστήρια. Έχουμε έναν άλλο κλάδο που είναι η ε, πιστοποίηση συμβουλευτική, ο άλλος κλάδος είναι ο συμβουλευτικός και της κατάρτισης και βέβαια ε, δεν χρειάζεται να σας διαβάσω ολόκληρη τη διαφάνεια. Θα έχουμε εξάλλου να κάνουμε με διάφορες ερωτήσεις σήμερα σχετικά με τον τομέα της ε, έγκρισης τύπου. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις στις Βρυξέλλες και στη Γενέβη, όπου είμαστε παρόντες ε, και συμμετέχουμε σε πολλές ομάδες εργασίας. Είναι μια από τι ιδιαιτερότητε της ε, ΟΤΑΚ, είναι ένα από τα ισχυρά μας σημεία, ότι δηλαδή συμβάλλουμε στην εμπειρογνωμοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε παρόντες σε σχετικέ ε, συζητήσει, διεθνεί ή ευρωπαϊκέ. Παγκόσμια διεθνή αναγνώριση και θα επιμείνω εδώ στο γεγονός ότι είμαστε τεχνική υπηρεσία για τη Γαλλία, για την Αγγλία, για τις κάτω χώρες και για τη Ρουμανία, με τέσσερις χώρες δηλαδή. Έχουμε διεθνείς ε, αναγνωρίσεις, αλλά που δεν είναι τόσο εντός θέματος σήμερα, για τις ε, δοκιμές και την εμπειρογνωμοσύνη. Εδώ έχουμε τα διάφορα εργαστήρια και κάνουμε τις ε, τυπικές και καθορισμένες δοκιμές. Ε, ξέχασα να σας πω, έχουμε, πέντε, έχουμε ένα εργαστήριο για ΟΝΚΑ ε, 4, Κάνουμε και σχέδια για δοκιμές, όταν έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη εντολή, με διαδοκιμές ε, σύγκρισης ε, ή επιδόσεων για συγκεκριμένα προϊόντα όταν αυτό μας ζητηθεί. Για τα εργαστήρια λοιπόν που και την εμπειρογνωμοσύνη παρά να σας πω πολλά θα σας δείξω τις διαφάνειες για να σας δείξω ότι έχουμε τα εργαστήριο περιβάλλοντος όπου γίνονται οι εργασίες για το θόρυβο, για τις δονήσεις, ε, τους κραδασμούς και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα καθώς και τις εκπομπές και την κατανάλωση με εργαστήρια τελευταίας τεχνολογίας. Ε, ε, για την ασφάλεια επίσης εργαζόμαστε για την ε, ενεργή και για την παθητική ασφάλεια αλλά και για ό,τι αφορά την αξιοπιστία. Και επειδή έχουμε δύο κέντρα δοκιμών έχουμε και πάρα πολλές πίστες για να μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε και να κυρώσουμε τις ε, επιδόσεις των τροχοφόρων, όλων των τροχοφόρων. Και τώρα, αν επιτρέπετε να δώσω το λόγο και άδελφο. Όχι, ε, θα περάσουμε πρώτα στην ερωτήσει. Σήμερα το πρωί είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο. Απόψε δεν θα έχουμε παραπάνω χρόνο, γι' αυτό και θα είμαι αυστηρή με το χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας. Να το γνωρίζετε το λέω, να σας ενημερώσω. Σάλμπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη μου ερώτηση είναι όταν εσείς ε, καταλάβατε ότι υπήρχε διαφορά εκπομπών ε, στα δοκιμές εργαστήριο και στις εκπομπές ε, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, τι κάνατε, κάνατε κάτι γι' αυτό. Oui, merci pour la σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όταν μιλάτε για εκπομπές, τι, για τι είδους εκπομπές μιλάτε, παρακαλώ. Τον έλεγχο εκπομπών, ανάλογα με το αν είναι συνθήκες εργαστηρίου ή πραγματικές συνθήκες. Καταλάβατε ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά, γιατί εδώ το ξέρουμε. Τι κάνατε γι' αυτό, κάνατε κάτι? Μιλάτε για τα οξύδια του αζώτου, κουμπέ οξυδίων του αζώτου. Μάλιστα. Ενημερωθήκαμε για αυτή την απόκληση όταν ε, είχαμε πρόσβαση στις ε, δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες με το νέο σύστημα RDE. Εμείς ε, ως τεχνική υπηρεσία δεν έχουμε εντολή να μελετήσουμε αυτές τις αποκλήσεις ως τεχνική υπηρεσία. Εμείς σήμερα εφαρμόζουμε την νομοθεσία που ισχύει, όπως αυτή περιλαμβάνεται στα ισχύοντα κείμενα. Εμείς λοιπόν παραμένουμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας και σήμερα η εφαρμόσιμη νομοθεσία, η ισχύουσα νομοθεσία και η μέτρηση των εκπομπών γίνεται μόνο στο εργαστήριο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια νέα πρόταση ώστε ο έλεγχος των εκπομπών να γίνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Πώς πιστεύετε ότι αυτό θα σας επηρεάσει ε, στις διαδικασίες που ακολουθείτε και δεύτερον πώς θα επηρεαστούν τα αυτοκίνητα και η τεχνολογία diesel. Γιατί η βάση θα είναι πολύ πιο απαιτητική. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν αυτές οι τεχνολογίες να προσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα ε, απέτηση και στην πραγματικότητα. Ναι, μάλιστα. Έχετε δίκιο ότι σήμερα με τη νέα νομοθεσία που υιοθετήθηκε το RDE θα έχουμε εκπομπές πολύ πιο κοντά με, σε αυτές που γίνονται στην πραγματικότητα γιατί θα μετρώνται οι εκπομπές ε, επιτόπου και όχι μέσα σε ένα εργαστήριο. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη των αυτοκινήτων θα είναι διαφορετική διότι θα υπάρχει πολύ πιο αυστηρό βαθμός ανοχής από ό,τι ισχύει σήμερα. Από αυτή την άποψη λοιπόν τα οχήματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις εκπομπές. Και Και βέβαια η εφαρμογή όλων αυτών θα ξεκινήσει μόνο από το 2019. Όσον αφορά την τεχνολογία, Υπάρχουν ήδη πολλές τεχνολογίες στην αγορά, αλλά θα πρέπει να ε, ενισχυθούν ώστε να μπορούν να λειτουργούν ε, υπό κάθε συνθήκη. Αυτό παίρνει ίσως κάποιο χρόνο, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες όπως το SR για το diesel, εφόσον μιλάμε για diesel, που είναι αποτελεσματικές. Πρέπει να δουλευτούν λοιπόν αυτές τις τεχνολογίες και να ενισχυθούν. Αυτό θα, στάλλο θα είναι υποχρεωτικό λόγω του ΕΡΔΕ. Είστε αισιόδοξοι δηλαδή, δεν νομίζετε ότι αυτό θα επιβάλλει κάποια ε, περιορισμού στη βιομηχανία του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. θα συνεχίσουν δηλαδή τα αυτοκίνητα diesel, μάλλον θα πρέπει τα αυτοκίνητα diesel να προσαρμοστούν στι νέε πιο απαιτητικές συνθήκε. Κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά τι τεχνικέ υπηρεσίε. περισσότερο είναι ερώτηση που αφορά του κατασκευαστέ αυτή που υποβάλλεται. Εμεί μπορούμε να πούμε μόνο πω για κάθε νέα νομοθεσία πρέπει να υπάρξει λίγο χρόνο για να μπορέσουν οι ε, κατασκευαστές αλλά και οι κατασκευαστές, αυτοκινήτων αλλά και αυτοί που κατασκευάζουν τους εξοπλισμούς των αυτοκινήτων να προσαρμοστούν ε, στο νέε απαιτήσει ώστε το RDE να μπορεί να εφαρμοστεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Γκερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δυο σας που είστε εδώ. Το iPad μου σβήνει μόνο του και δεν λειτουργεί μετά και το δακτυλικό μου αποτύπωμα. Λοιπόν, Ευχαριστώ πολύ για τις ειλικρινείς απαντήσεις σας, για το κατά πόσον ε, τα παράθυρα ε, ε θερμοκρασίας και ή ε, το σβήσιμο του, των διατάξεων μετά από 20 λεπτά αποτελούν διατάξεις αναστολής ή όχι. και επίσης για το ότι θεωρείται πως η συνήθιση χρήση είναι χρήση εκτός εργαστηρίου για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς μπορούμε να δοκιμάζουμε αυτοκίνητα πέραν του συνήθους κύκλου ε, NEDC. Λέτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχετε τη δυνατότητα συστηματικά να εντοπίζουμε διάταξη, διατάξεις αναστολής με βάση τον, τους ισχύοντες κανονισμούς. Είναι η απάντηση στην ερώτηση 8. Γιατί όχι, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε υπό την προπόθεση ότι δεν το χρησιμοποιείτε με, για την επίσημη έγκριση τύπου. Μπορείτε όμως να το χρησιμοποιήσετε λέγοντας τον κατασκευαστή, ε, ρωτώντας τον γιατί είναι 20 φορές περισσότερο μεγαλύτερες οι εκπομπές να χρησιμοποιήσουμε άλλου τύπου κύκλο. Επίσης, αλλάζοντας το λίγο ή γυρίζοντας το ανάποδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα ακόμα και μέσα στο NDC. Καταλαβαίνω ότι επίσημα δεν μπορείτε να το κάνετε, αλλά μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διασταυρώσετε τα αποτελέσματα του NDC με αποτελέσματα άλλων κύκλων που μπορείτε εσείς να χρησιμοποιήσετε στα εργαστήρια. Γιατί δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνατε στο παρελθόν. Merci beaucoup. Ναι, ε, πολύ κέρια η ερώτησή σας. Το είπατε και εσείς θέτοντας την ερώτηση. Από νομικής πλευράς ως τεχνική υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε την νομοθεσία ε, που είναι ισχύ για όλους σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δηλαδή ως τεχνική υπηρεσία στη Γαλλία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από την τεχνική υπηρεσία της Ισπανίας κλπ. Γιατί αλλιώς θα είχαμε στρεβλώσεις ε, απαραδεκτές. Δεν θα είχαμε και πολλούς πελάτες αν το κάναμε, <laughs> για να είμαι πολύ ειλικρινής. Τώρα, αν μας το ζητήσουν οι αρχές, μάλλον ε, αν μα το ζητήσουν οι αρχέ, θα μπορούσαμε να το, ζητούσαν οι αρχές θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλά θα είμαι και πάλι ειλικρινή. αυτό έχει ένα κόστος και δεν πληρωνόμαστε για να ε, κάνουμε τέτοιου είδου δοκιμές κάνουμε δοκιμές έγκριση τύπου όπω αυτές προβλέπονται από τον νόμο και από τους κανόνες τίποτα παραπάνω ε, ερώτηση Καμία εθνική αρχή δεν σας το ζήτησε ως τώρα, έτσι δεν είναι. Ε, παρ' όλα αυτά είναι νομική τους υποχρέωση να εφαρμόζουν ε, την ε, ε, κοινοτική νομοθεσία. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αναφέρεται στις διατάξεις αναστολής και έχουμε δει και πολλές μελέτες και άλλα στοιχεία που υποδεικνύουν ε, αποδεικνύουν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γνώριζαν, συνειδητοποιούσαν ότι χρησιμοποιούνται διατάξεις αναστολής προκειμένου να υπερκεραστούν ε, ε, οι δοκιμές. Εσείς ποτέ δεν χρησιμοποιήσατε κανένα, καμία άλλη δοκιμή εκτός από την NEDC. Απάντηση. Και πάλι να σας πω ότι ποτέ δεν μας ζητήθηκε σε, στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου να ζητήσουμε ε, τι συμβαίνει ε, για θέματα τα οποία ε, ξεπερνούν τις, τις δοκιμές οι οποίες προβλέπονται. Εσείς για τον εαυτό σας από περιέργεια δεν το κάνατε ποτέ. Όχι. Ε, ένα Σάββατο πρωί, ένα Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο λέει η κυρία Λόπε. Όχι, ειλικρινά. Ε, ποτέ δεν κάνουμε οποιαδήποτε πειραματισμό εκτός του κύκλου. Θα προεκτείνω τις προηγούμενες ερωτήσεις. Η, Βασιλική Επιτροπή, την οποία δημιούργησε ε, η υπουργό ε, ε, σας ζήτησε να εξετάσετε 85 οχήματα μέσω της χρήσης συσκευών PEMS, φορητών συσκευών μέτρησης καυσαερίων μπορείτε να μας πείτε, να μας δώσετε μια ιδέα για τα αποτέλεσματα που προέκυψαν και πώς έγινε αυτό το πείραμα. Ναι, ε, πράγματι η ε, Βασιλική Επιτροπή όπως ονομάστηκε ε, μας ανέθεσε να κάνουμε αυτές τις δοκιμές. Κάναμε τριών τύπων δοκιμές. Πρώτον, D1, έτσι την ονομάσαμε. η δοκιμή αυτή Ε, ε, προσπαθήσα, ε, είχε ως ε, στόχο να δούμε αν το, το όχημα αντιλαμβανόταν ότι βρισκόταν στο εργαστήριο στην αρχή, σε ένα κίνημα νοημάντα. Δεύτερον, αλλάξαμε τα αρχικά settings και είδαμε, προσπαθήσαμε να δούμε αν υπάρχουν διαφορές. Και τρίτον, ε, τοποθετήσαμε μια φορητή συσκευή σε ένα PEMS, ε, σε, κανονικές, ε, συνθήκες ε, και προσπαθήσαμε να αναπαράγουμε τον κύκλο NEDC. Με αυτές τις τρεις δοκιμές, οι οποίες ξεπερνούν το όριο το, τον, της ε, νομοθεσίας προφανώς, ε, ε των υποχρεώσεων που μας επιβάλλει η νομοθεσία, είδαμε διαφορές. Ε, είπατε ότι ξεπερνούν το όριο της νομοθεσίας. Όμως στην νομοθεσία λέει, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ρητά ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τη χάνουν σεβασμού σε κανονικές συνθήκες. Ε, πολλοί Πήραμε πολλές απαντήσεις ε, για το τι είναι αυτέ οι κανονικέ ε, συνθήκες. Εμείς θεωρούμε ότι οι κανονικέ συνθήκες δεν είναι αυτές του εργαστηρίου. Με βάση τα αποτελέσματα τα δικά σα που δημοσιεύθηκαν και είναι διαφανή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες, πολύ σημαντικέ ε, διαφορές, αποκλήσει ανάμεσα στις πραγματικές εκπομπέ και τι εκπομπέ των δοκιμών του εργαστηρίου. Πήρατε μέτρα πήρατε τα μέτρα που θα έπρεπε ή να αποσύρετε, να ανακαλέσετε δηλαδή τις εγκρίσεις τύπου ή να προβείτε σε πρόσθετες έρευνες. Ε, η απάντηση είναι σαφέστατη. Εμείς είμαστε τεχνική υπηρεσία μόνο, τίποτα άλλο. Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την υποβάλλετε στις γαλλικές αρχές. Ε, δεν μπορούμε εμείς να αποσύρουμε μια έγκριση τύπου. Κάνατε προτάσεις, υποδείξεις στις ε, γαλλικές αρχές για το τι θα έπρεπε να κάνουν. Ε, αναφέρατε την Βασιλική Επιτροπή, συγγνώμη, την Επιτροπή Ρουαγιάλ, συγγνώμη. Ε, ε, κατόπιν των, των δοκιμών μας προέκυψαν εκεί διάφορα πορίσματα τα οποία προφανώς βαίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. επόμενη ερώτηση ε, αναφερόμαστε, ε, έχουμε μιλήσει για τα ε, θερμικά παράθυρα ε, και άλλες διατάξεις, οι οποίες φαίνεται να είναι διατάξεις αναστολής. Τη σχολιάσατε. εμείς με τη ΦΙΑ δεν έχουμε ασχοληθεί, οπότε τις διατάξεις ΦΙΑ δεν τις έχουμε δει ποτέ. Τα θερμικά παράθυρα τα έχουμε δει, όχι όμως σε... Τα γνωρίζουμε, αλλά όχι στο πλαίσιο της ε, έγκρισης τύπου. Δεν μιλούσα για έγκριση τύπου, μιλούσα για, την, για τις ε, δοκιμές στα 85 αυτοκίνητα. Ναι, πράγματι, εκεί είδαμε διαφορές. Και ο κατασκευαστής μας εξήγησε για ποιο λόγο υπήρχαν αυτές οι, οι διαφορές, αυτές οι αποκλήσεις. Ε, πώς θα σας φαινόταν η, ιδέα μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ε, πάνω από τις εθνικές ε, ε, υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσουμε το σύστημα θα είναι πιο αποτελεσματικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι καλή ιδέα. Απάντηση. Ε, ε, δεν μιλώ βέβαια εκ μέρους των γαλλικών αρχών. Εμείς ως εταιρεία ε, ειλικρινά θα θέλαμε να υφίσταται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου έτσι ώστε όλες οι τεχνικές υπηρεσίες να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο. Το ζητάμε, το επιθυμούμε, προκειμένου να αποφεύγουμε διαφορετικές ερμηνείες α, μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών. Έτσι ώστε οι κατασκευαστές να μας λένε «Ξέρετε κάτι, ο διπλανός κάνει κάτι διαφορετικό, εσείς δεν το κάνετε» κλπ. Θα θέλαμε λοιπόν ε, μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου. Συγγνώμη που σας, δεν σας προηγουμένω. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω να κάνω για να διευκρινίσω κάτι, κάποια πράγματα. Η οργάνωσή σας είναι σε τεχνικό μόνο επίπεδο ή είσαστε και η αρχή η οποία χορηγεί τι εγκρίσει τύπου. Εμεί είμαστε η τεχνική υπηρεσία και αυτό περιλαμβάνει πολλά πράγματα και η γαλλική αρχή η οποία δίνει την έγκριση τύπου ονομάζεται CNRV το CNRV λοιπόν υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε τέτοια δημόσια αρχή. Μάλιστα. Άρα η ερώτησή μου και νομίζω ότι αυτό αναρωτιούνται και οι συνάδελφοι μετά από αυτά που ακούσαμε και από τους άλλους προσκεκλημένους σήμερα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον, σε ό,τι αφορά και τις διατάξεις αναστολής και τα λοιπά που συζήτησαν οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, λοιπόν, είναι σημαντικό ότι εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να καταλάβουμε τι θα πρέπει να βελτιώσουμε στο σύστημα προκειμένου να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την παραπλάνηση από πλευρά των παραγωγών προς τους καταναλωτές σε σχέση με τα αυτοκίνητα που αγοράζουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των OEM που πληρώνουν για την έγκριση τύπου, άρα θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία και ενδεχομένως να υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων. Πώς μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν το σύστημα στην Ευρώπη και πώς θα μπορούσε να διοργανωθεί και κάτι σε διεθνικό επίπεδο αυτό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επιλύσει κάποια προβλήματα ή πιστεύετε ότι θα σαν πιο μικρές αναπέστατες αλλαγές. Και σας δίνω τα υπόλοιπα τρία λεπτά μου για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω. Αυτό που είδαμε τον τελευταίο χρόνο είναι το εξής, ότι η έγκριση τύπου δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις διαστάσεις και έτσι υπάρχουν κάποια οχήματα τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία δεν είχαμε εντοπίσει. Με πάσα ειλικρίνεια. Θεωρώ ότι η παρακολούθηση υποπτή της αγοράς θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες που εκφράζονται. Γιατί Εκεί είναι η πραγματική λειτουργία του οχήματο. Δεν ξέρω αν αυτέ είναι οι φυσιολογικέ συνθήκε λειτουργία. Αυτό εξαρτάται φυσικά και σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του οδηγού. Αλλά θεωρώ ότι η υποπτία τη αγορά θα αρκούσε. Τώρα, κατά πόσο να θα οργανώνονταν σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση στην ερώτηση που θέσατε. Μάλιστα. Άρα η υποπτία τη αγορά η παρακολούθηση της αγοράς θα είχε να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται το όχημα στον πραγματικό κόσμο μετά την πώλησή του. Αυτό θεωρώ ότι ρώτησε και ο συνάδελφος Γερμπράντη προηγουμένω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι νομικές προδιαγραφές και είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις νομικές διατάξεις και να γίνονται αντιστοίχω και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι το εξή. Μία οργάνωση πώς η δική Γιατί δεν θέτει πιο βασικά θεμελιώδη ερωτήματα. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι, για παράδειγμα, έχει νόημα αυτό που ζητάει ο νόμος. Στην ιατρική, για παράδειγμα, οι γιατροί υποχρεούνται να συμπληρώνουν έντυπα και διάφορα έγγραφα που δεν έχουν να κάνουν με τους ε, ασθενείς απαραίτητα. Αλλά ως γιατροί, για παράδειγμα, ξέρουν κάτι παραπάνω για τους ασθενείς. Εσείς αντίστοιχα, γιατί δεν κάνατε ε, προτάσεις για τις, πώς να βελτιωθεί η νομοθεσία και γιατί δεν το κάνετε αυτά τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, η απάντησή μου θα είναι μάλλον άμεση. Σήμερα οι κανόνες διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και αν ένας καλός ε, γιατρός ε, για παράδειγμα, έχει μια διέστηση. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε, κοιτάξτε κύριε κατασκευαστή, ε, έλατε εδώ και δεν πειράζει, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Όχι, εμάς μας πληρώνουμε για να κάνουμε τις συγκεκριμένες δοκιμές, τα συγκεκριμένα τεστ. Είτε θα μας δώσει μια σαφή αρμοδιότητα η νομοθεσία για να κάνουμε αυτοσχεδιασμούς αυτό θα ήταν μια διαφορετική διάσταση. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έρευνα. Έτσι όπως έχει σήμερα η νομοθεσία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τέτοιο. Και θα ήθελα να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι η μελλοντική νομοθεσία σε ό,τι αφορά το RDE, τα επίπεδα θερμοκρασίας και το καθεξής, θεωρώ ότι αυτά ενισχύουν την κατάσταση. Δηλαδή, αν περάσει ένα όχημα όλα αυτά τα τεστ, είναι πραγματικά πολύ στενερό και μετά θα πρέπει να εγκριθεί και να επιβεβαιωθεί η κατασκευή κτλ. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Ζανόφσκι έχει το λόγο. Mm. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, τα τεστ αυτά, τα OEC, τα EDAC, Προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο, δεν είχατε την αίσθηση ότι κάτι περίεργο γινόταν, ότι κάτι ελόχευε. ότι ενδεχομένω και να χρησιμοποιούνταν δηλαδή διατάξει ανάστολη κατά τη διάρκεια των τεστ, των δοκιμών που διεξάγατε. Δεν είχατε κάποια διέστηση, δηλαδή ότι κάτι στραβά πήγαινε. Ε, με απόλυτη ειλικρίνη σας απαντώ πως όχι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Στην απάντησή σας στην ερώτηση παριθμών 8 αναφέρεται ότι σήμερα με την τρέχουσα νομοθεσία και τους τρέχοντες κανόνους δεν είστε σε θέση να εντοπίσετε παράνομες διατάξεις αναστολής. Πιστεύετε ότι η νέα πρόταση που χρησιμοποιείται το σύστημα RDE επιλύει το πρόβλημα αυτό. για την δοκιμή και για την έγκριση του τύπου. Το νέο σύστημα σας δίνει επαρκή εργαλεία ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο επιπλέον πέρα από αυτά που προβλέπονται. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις ε, αναστολής όντως ε, τα μελλοντικά κείμενα, η μελλοντική νομοθεσία θα καλύψει πολύ πιο πολλές διατάξει Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία θα τεθούν όρια πολύ πιο ευρεία σε σχέση με τις δοκιμές στο εργαστήριο και αυτό σαφώς θα μας βοηθήσει. Από την άλλη, το να εντοπιστούν παράνομα ή νόμιμα στοιχεία εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Γιατί αυτό είναι και θέμα λογισμικού. Και σήμερα δεν προβλέπεται τίποτα τέτοιο στο κείμενο. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Τελευταία ερώτηση. Σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών έγινε μία συζήτηση για την έγκριση συστημάτων οχημάτων και εξετάσαμε μια ενδεχόμενη υπηρεσία εποπτείας η οποία θα παρακολουθεί τέτοιου είδους μηχανισμούς. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιπλέον ουραφιοκρατία. ένα επιπλέον ε, επίπεδο παρακολούθησης ενδεχομένω να μην μας οδηγήσει σε οποιαδήποτε λύση. Το θέμα θα ήταν να υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες ή ένα σύστημα ελέγχου το οποίο θα αξιοποιούσε την τελευταία τεχνολογία, την ε, τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μία επιπλέον αρχή παρακολούθησης ουσιαστικά θα έχει Ω αποτέλεσμα επιβάρυνση με επιπλέον γραφειοκρατία. Δεν φοβάστε λοιπόν την επιπλέον αυτή η διάσταση τη γραφειοκρατίας. Ναι, όντω. Αν τελικά το αποτέλεσμα είναι πιο πολύ γραφειοκρατία, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει σε τίποτε. Εμείς ναι, ως τεχνική υπηρεσία, αυτό που θέλουμε είναι να είναι ταυτόσιμη για όλους η ερμηνεία της νομοθεσίας. Ή αν θα μπορούσε να υπάρχει μία υπηρεσία η οποία θα ελέγχει ότι όλες οι αρχές εφαρμόζουν με τον ίδιο τρόπο α, την νομοθεσία, αυτό θα μας βοηθούσε ήδη πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα προσθέτεται γραφειοκρατία ή όχι. Κοιτάξτε, σήμερα δεν έχουμε απάντηση να δώσουμε στο θέμα του λογισμικού για την ανείχνευση τέτοιων διδάξεων. Δεν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Ο κύριο Γερμπράντη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Μία πολύ απλή ερώτηση, διευκρινιστική, επιτρέψτε μου. Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ε, μία λίστα των εθνικών αρχών αναχώρα για την πιστοποίηση και στην Γαλλία αναφέρεται για τα μηχανοκίνητα οχήματα διρεξιών Technique UDAC. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η δική σας εταιρεία. Σας ε, αναφέρουν λοιπόν στην ιστοσελίδα ως Εθνική Αρχή για Παρακολούθηση της Αγοράς. Αυτό τι σημαίνει ότι πέρα από την τεχνική υπηρεσία που παρέχετε, διαδραματίζεται και ρόλο ως αρχή παρακολούθησης και υποπτίας. Απάντηση. Κοιτάξτε, είναι λάθος. Λάθος. Σφάλμα. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση η αρμόδια αρχή εποπτείας στη Γαλλία. Μάλιστα. Ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε. Άλλη ερώτηση. Τι προτίθεστε να κάνετε εκτός των τεστ ε, EDC που περιγράφονται. Αν και παράδειγμα οι γαλλικές αρχές σας ζητούσαν να δοκιμάσετε να κάνετε έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο με πολύ διαφορετικούς τρόπους πέρα από το standard test NEDC θα μπορούσατε και θα θέλετε να αναλάβετε την, το καθήκον αυτό. Οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ζητούν ε, την εκτέλεση ελέγχων για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο, για τη διάσταση της ασφάλειας κτλ. Αν προς το σκοπό αυτό ζητηθούν επιπλέον έλεγχοι, μπορούν να το ζητήσουν και θα τις εκτελέσουμε τους ε, ελέγχους αυτούς. Και αυτό έγινε λοιπόν ε, και στην περίπτωση της Επιτροπής Ρουαγιάλου. Μάλιστα, λέει ο κ. Γεμπράντη, γιατί σε μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις είπατε ότι δεν είστε σε θέση να το κάνετε αυτό ως τεχνική υπηρεσία, γιατί υπάρχει και ο ανταγωνισμός με τους άλλους. Αλλά θα μπορούσατε να κάνετε τέτοιο έλεγχο αν σας ζητηθεί. Κοιτάξτε, η απάντηση που έδωσε προηγουμένως είχε να κάνει σε ένα συστηματικό επίπεδο. Δεν γίνεται αυτό να το κάνουμε δηλαδή για κάθε έγκριση τύπου γιατί προβλέπεται από την νομοθεσία σε ό,τι αφορά το NEDC. Τώρα, φυσικά, αν μας το αναθέσει οι αρχές, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε περίπτωση που ισχύουν διαφορετικοί όροι και συνθήκε πέρα από τι συνθήκε για τη χορήγηση έγκριση τύπου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, τώρα σε ό,τι αφορά το μέλλον, γιατί αυτό ασφαλώ είναι το άλλο σκέλο. Ένα πράγμα που μα απασχολεί εδώ στην Επιτροπή είναι η ανταγωνιστικότητα, ο ανταγωνισμό μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και των αρχών χορήγηση έγκριση τύπου θεωρείτε ότι ο ανταγωνισμός αυτός είναι υγιής, είναι μια υγιής έτσι άμυλα ή είναι κάτι που θα έπρεπε στο μέλλον να φροντίσουμε να κατασταλεί. Απάντηση. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση είναι ο ανταγωνισμός για την ερμηνεία των κανονισμών. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός να ευνοεί κάποιον, κάποια τεχνική υπηρεσία πιο πολύ από ότι κάποια άλλη, για να είναι δηλαδή πιο ευνοϊκή σε ό,τι αφορά την εκτέλεση ε, των ελέγχων. Αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να Μάλιστα. Αλλά αυτό που παρατηρούμε επίσης είναι ότι υπάρχει και μια τάση στα κρατημέλη πώς να σας το πω, πώς να το διατυπώσω με τον σωστό τρόπο. Διακρίνουμε μία τάση να υπάρχει μία χαλαρότητα ενδεχομένως κάθε χώρα να βοηθάει την εθνική της βιομηχανία να περάσει τον νόμο και τις νομικές εντάξεις. Δεν λέω ότι είναι παράνομο αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια αμοιβαία συμφέροντα προφανώς σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου κάποιων οχημάτων έχετε την αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν μιλάω μόνο στη Γαλλία. Στην Ιταλία, σε άλλες χώρες, έχετε την αίσθηση από τη δική σας εμπειρία και από τη δική σας γνώση ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απάντηση. Κοιτάξτε, να σας πω για τη Γαλλία. Δεν μπορώ να σας πω τι γίνεται αλλού, αλλά να σας εγγυηθώ ότι στη Γαλλία η ερμηνεία είναι πολύ στεναρή και αυστηρή. δεν υπάρχει αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση μεταξύ των αρχών και των κατασκευαστών. Δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε για κάποια άλλη αρχή, για κάποια άλλη χώρα. Κυρία Κόνισνα. Eh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Έχω μια-δυο ερωτήσεις ε, και σε σχέση με τις ερω... γραπτές απαντήσεις που μας στείλατε. Στην ερώτηση υπάρχουν 8 λέτε ότι τα θέματα που συνθέεται με τις συσκευές αναστολής μπορέσατε να ενημερώσετε την Κομισιόν για αυτά και έπειτα εξετάσατε την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ποια συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιήσατε και ποιο ήταν παρόν από πλευρά τη Κομισιόν, πότε του ενημερώσατε, σε ποια συνεδρίαση. Oui, alors je, voudrais juste apporter une petite correction. Donc... Θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση. Όντω, εγώ είχα λάθο ερμηνεύσει το δεύτερο τμήμα. Όταν απαντήσαμε ότι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε διάφορε ομάδε εργασία, αυτό αφορά το γεγονό ότι ω τεχνική υπηρεσία είμαστε υπέρ οδηγών για μια μεθοδολογία. Ε, οπότε εγώ το κατάλαβα ότι με ρωτήσατε κατά πόσο αυτή μας η βούληση εκφράστηκε στην Κομισιόν. Εμείς λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές στην Κομισιόν ότι ως τεχνική υπηρεσία είμαστε υπέρ της ε, δημιουργίας διαδικασιών όπου δεν θα χωράει ερμηνεία διαφορετική από κάθε ε, τεχνική υπηρεσία. Λυπούμε, είναι δικό μου λάθος, λάθος κατάλαβα. Μάλιστα. Ωστόσο, να σας ρωτήσω, με ποιον συζητήσατε στην Κομισιόν, πότε ήταν περίπου αυτή η συνεδρίαση που θέλατε να τους ενημερώσετε ότι θέλετε διαφορετική διαδικασία, γιατί αυτή η διαδικασία δεν είναι τέλεια. Παρακολουθούμε εδώ και 30 χρόνια και πάνω την σχετική ομάδα εργασία. Τώρα να σα πω σε ποια συνεδρία είπαμε ότι ναι, θέλουμε να έχουμε ξεκάθαρου κανόνε. Δεν μπορώ για να σα το πω με ακρίβεια. Από τη δεκαετία του 70 έχει ξεκινήσει αυτή η δουλειά. Είχαμε και τότε την πρώτη οδηγία για μέτρηση των εκπομπών. Από τότε συμμετέχουμε στην εκπόνηση νομοθε... της νομοθεσίας. Σε αυτή τη τεχνική ομάδα εργασίας, όπου είναι ένας κόσμος, όπου καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα, εμείς ως τεχνική υπηρεσία θέλουμε ξεκάθαρες διαδικασίες πιστοποίησης, έγκρισης τύπου. Είναι προς το συμφέρον μας να, τονίσουμε, να το τονίσουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα δεν είμαι εγώ εκεί εδώ και 40 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι σαφές ότι είναι προς το δικό μας συμφέρον να έχουμε ξεκάθαρες διαδικασίες και προ αυτή την κατεύθυνση απαντήσαμε ότι όντω έχουμε ενημερώσει την Κομισιόν για αυτή μας την ε, βούληση και επιθυμία. Λέτε πόσο δύσκολο είναι να οριστεί η φυσιολογική χρήση. Εσείς τι ορισμό έχετε να προτείνετε. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Είναι περίπλοκο γιατί Παρακολουθήσαμε από κοντά την εκπόνηση του κανονισμού ΕΡΔΕ και μπορώ να σας πω ότι ώρες επί ώρων συζητήσαμε για να καταλήξουμε στις ε, οριακές συνθήκες. Ε, τώρα τι είναι μια φυσιολογική κατάσταση οι φυσιολογικές συνθήκες είναι στα Βόρεια Ευρώπη, είναι στη Νότια Ευρώπη, ανατολικά, δυτικά, σε ποιο υψόμετρο, σε ποια θερμοκρασία. Υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές χρήσεις που δεν είναι καθόλου εύκολο να ορίσουμε τι είναι η φυσιολογική χρήση. Στο RDE λοιπόν υπάρχουν ορισμοί όπου μπορούμε περισσότερο να βασιστούμε, αλλά ειλικρινά δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και θέλω να συνεχίσω για αυτή την υπόθεση της φυσιολογικής χρήσης γιατί στην ερώτηση 10 λέτε ότι για την φυσιολογική χρήση είναι έλλειψη του κανονισμού το να μην ορίζεται η φυσιολογική χρήση. Εσείς έχετε ενημερώσει κάποιον, γιατί τώρα λέτε πως είναι πρόβλημα, αλλά ο, ο, ο νομοθεσία αυτή ισχύει εδώ και δεκαετίες. Φαντάζομαι ότι σε κάποιον θα το έχετε πει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μελετήσει πραγματικά αυτό το κομμάτι, διότι είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια πριν να εγκριθεί το RDE, ναι, αλλά εγώ δεν σας ρωτάω αν το μελετήσατε, αλλά αν διαπιστώσατε ότι δεν είναι σαφής ο ορισμός και ότι άρα θέλετε να ενημερώσετε. Ναι, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι μέχρι στιγμής οι εκπομπές και οι διαδικασίες έγκρισης τύπου γίνονταν στα εργαστήρια. Οπότε για... εκεί δεν χρειαζόμαστε τον ορισμό της ε, ε, φυσιολογικής χρήσης. Τώρα περνάμε σε μια άλλη διάσταση με το ΑΡΔΕ και εκεί τίθεται το θέμα για τη, φυσι... τη φυσιολογική χρήση. Μέχρι σήμερα δεν χρειαστήκαμε τέτοιον ορισμό. Ενδιαφέρουσα αυτή η δήλωση, διότι από όσο γνωρίζουμε τα αυτοκίνητα πρέπει να συμμορφούνται προς την νομοθεσία και στο ε, λέει ε, όρια εκπομπών για φυσιολογική χρήση. Ε, για, μας, για σας αυτό σημαίνει εκτός εργαστηρίου. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει το NDC για την έγκριση τύπου, αλλά επίσης η ίδια νομοθεσία λέει ότι πρέπει να τηρείται ένα συγκεκριμένο όριο εκπομπών και για παράδειγμα ότι οι συσκευέ αναστολή απαγορεύονται. Και αυτά πρέπει κανεί να τα ελέγξει, γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σύμμορφο προ την νομοθεσία. Στην προηγούμενη σα απάντηση είπατε ότι ποτέ δεν σα απασχόλησε να εξετάσετε αυτά τα θέματα. Και είπατε ότι στι δοκιμέ είναι δύσκολο διότι δεν υπάρχουν κανόνε για κάτι τέτοιο. Όμω πώ μπορεί να υπάρχουν λεπτομέρειε κανόνε, α πούμε για την αναγνώριση ή τον εντοπισμό μιας τέτοια συσκευή, γιατί αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό κάθε αυτοκίνητο. Αν όμω εσεί σκεφτείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα κάνετε δοκιμέ παραπάνω. Γιατί δεν κάνατε. Κοιτάξτε, για να δούμε αν κάτι δεν είναι φυσιολογικό, εάν αυτό γίνεται δηλαδή σε ένα πλαίσιο defeat device, ε, πρέπει να το ψάξουμε. Γιατί αν εφαρμόσουμε την νομοθεσία όπως έχει τώρα, στους, ανάμεσα στους 20 και τους 30 βαθμούς, δεν θα ψάξουμε τι θα γίνει ε, σε ψηλότερη ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Έτσι όπως ήταν η νομοθεσία λοιπόν πριν το RDE, ε, ε, οι δοκιμές γίνονταν ανάμεσα σε θερμοκρασία ανάμεσα στους 20 και τους 30 βαθμούς. Εάν δεν ψάξουμε τι γίνεται πριν ή μετά, πώς θα εντοπίσουμε την, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συσκευής. Καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσατε να το εντοπίσετε όταν κάνετε το RDE ε, για την έγκριση τύπου, αλλά όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι στον κόσμο ε, που κάνουν άλλες δοκιμές και έχουν διαπιστώσει ότι ένα ρενό, για παράδειγμα λέω, ε, έχει αδιαφορετικές επιδόσεις εκτός του θερμικού παραθύρου. Δεν σκεφτήκατε να κοιτάξετε κι εσείς λίγο πιο έξω για να, γιατί τα αυτοκίνητα πρέπει να συμμορφώνονται και στα περιβαλλοντικά στάνταρτ. Ε, έχετε δίκιο. Αυτό που σημαίνει στη Γαλλία σήμερα είναι ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστό ε, πως ε, οι εκπομπές δεν είναι εντάξει κάτω από 20 πάνω από 30 βαθμούς στη Γαλλία έχουμε αναλάβει δράση προκειμένου να διορθώσουμε αυτό το θερμικό παράθυρο που είναι πολύ στενό. Ωραία, για να δούμε, στην, να έρθω στην Επιτροπή Ρογιάλ. Εσείς εξετάσατε 86 μοντέλα, εσείς έτσι δεν είναι, ωραία. Ε, στην έκθεση αναφέρεται ότι το Renault Captur φάνηκε ότι υπήρχε λογισμικό παγίδευση οξυδίων του αζότου. Ε, αυτό ήταν στα πορίσματα, αλλά όχι στην τελική έκθεση. Είναι αλήθεια ότι βρήκατε παρατυπίες στο Renault Capture που ε, οδηγούσαν στο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει παγίδα οξυδίου του αζότου. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα ε, την οτσή σας. Ε, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στο Financial Times. Πρέπει να το διαβάσατε, δεν μπορεί. το θέμα της βαθμονόμησης στα Renault, αυτό εννοείται. Ήταν ένα άρθρο για την έρευνα στη Γαλλία όπου έλεγε το εξής. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε ε, δεν συμπεριέλαβε ορισμένο δυνερά συμπεράσματα γιατί την έκθεση την συνέταξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ε, όμως κάποιοι στην Επιτροπή σας είχαν πει φαίνεται ότι για το Renault Καπτύρι υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι χρησιμοποιείται ως software. Ε, όμως αυτό δεν συμπεριελήφθη στην τελική έκθεση. Ε, αν όμως ε, υπήρχε τέτοιο πόρισμα θα πρέπει να προήλθε από τη δική σας έκθεση. Όχι, εμείς δεν κάναμε ε, εμείς, εμείς ε, μετρήσεις για το software. Το κάτι κάνει μια άλλη εταιρεία. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά αν βλέπετε παράξενη συμπεριφορά, ε, την οποία μπορείτε να την αποδώσετε και να την εξηγήσετε μόνο με την ύπαρξη ε, λογισμικού, προφανώς αυτό προκύπτει από τις δικές σας δοκιμές. Απάντηση. Εμείς είμαστε εργαστήριο δοκιμών. Κάνουμε τις δοκιμές όπως μας τις ζητούν. το λογισμικό δεν είναι της αρμοδιότητάς μας. Της αρμοδιότητάς μας. Η Επιτροπή αυτή είχε ως στόχο πράγματι να διαλευκάνει και να διαφωτίσει όλες τις ε, παρατυπίες ή τις ανομαλίες που προκύπτουν ε, στα αυτοκίνητα που διακινούνται στη Γαλλία. Αυτό είναι το, αυτή είναι η αποστολή της Επιτροπής. Ε, τις ερωτήσεις αυτές πρέπει να τις υποβάλλετε στις αρχές. Εμείς κάναμε απλώς τις δοκιμές 86 μοντέλων, τίποτα άλλο. Εκεί σταμάτησε η εργασία μας. Κυρία Γκρουστέτ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και τις απαντήσεις σας. Θέλω να σας υποβάλω ένα πολύ απλό ερώτημα. Πότε μάθατε πότε συνειδητοποίησατε τις διαφορές ανάμεσα στις εκπομπές του εργαστηρίου και στις ε, εκπομπές σε κανονικές συνθήκες. Πότε ακριβώς συνειδητοποίησατε αυτή τη διαφορά, τις αποκλήσεις. Νομίζω μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Όταν δημοσιεύθηκαν κάποια άρθρα που ανέφεραν μετρήσεις με φορητές συσκευές, PEMS, που έδειχναν πως οι εκπομπές δεν ήταν ίδιες με αυτές του εργαστηρίου ερώτηση. Οπότε δεν είχατε ενδείξεις που να σας επιτρέπουν να φανταστείτε πως ε, πράγματι υπήρχαν διαφορές και αποκλήσεις. Και ποιες ήταν οι σχέσεις με τους ε, κατασκευαστές. Ε, σας, ε, είσαστε ανεξάρτητοι τελείως ή οι κατασκευαστές ε, σας δίνουν έτοιμα αποτελέσματα. Ποιες είναι οι σχέσεις σας μαζί τους. Πολλές ερωτήσεις μου υποβάλλετε. Ε, ε, είναι πασίγνωστο πλέον ότι η, η, παλιότερα η διαδικασία ήταν τέτοια που συμπεριλάμβανε πηγές βελτιστοποίησης. Δηλαδή είχε αντοχές ε, που ανάλογα με τις επιλογές που γινόντουσαν ε, μπορούσαν να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα. Ε, βελτιστοποίηση. Αυτές οι βελτιστοποιήσεις όμως ήταν νόμιμες. Όμως επουδενή δεν πιεστήκαμε ποτέ από κατασκευαστές προκειμένου να κάνουμε τις δοκιμές με τον α ή τον β τρόπο. Ε, η, τα περιθώρια ελαστικότητας που υπήρχαν, ε, ναι, χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές κατά το δοκούν, αλλά νομίμως. Ε, πράγματι μας μας πληρώνουν οι, οι, κατασκευαστές αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί. Ε, εδώ και 50 χρόνια αυτό κάνουμε και αν δεν ήμασταν ανεξάρτητοι δεν θα είχαμε επιβιώσει. Δεν έχουμε κανένα λόγο να χάσουμε αυτές τις αξίες. Ε, όχι, όχι. Ε, δεν ήταν η πόνη υποψία αυτό που εξέφρασα. Ήθελα απλώς να δω πώς είναι η σχέση με τους κατασκευαστές. Αυτό να μάθω. Για το μέλλον τώρα. Φαντάζομαι ότι υποχρεωθήκατε να κάνετε κάποιες τροποποίησεις για να εφαρμόσετε τον καινούριο κύκλο ε, οδήγηση ε, στον δρόμο. Ε, τι σημαίνει αυτό πλευρά οικονομικής για σας, επενδύσεων κλπ. Κυρία Γκροστέτ, έχετε και τα δύο time slots μαζί και... Όχι. Σταματάτε εδώ. Ε, πράγματι χρειάζεται να κάνουμε επενδύσεις για τον ε, WLTP που είναι ο μελλοντικό κύκλος αυτό ήδη το έχουμε ξεκινήσει και είναι σημαντικές επενδύσεις αυτές ενώ για το RDE ε, το Road Driving Emissions και εδώ έχουμε η επένδυση είναι 200-300 ευρώ για κάθε διάταξη PEMS, για κάθε συσκευή PEMS. Ε, βέβαια αυτό είναι για την αγορά μόνο, χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, είναι κάτι καινούριο, θα πρέπει να γίνει μια ολόκληρη δουλειά ε, προκατακτική, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σωστά οι συσκευές PEMS. Ε, όλα αυτά βέβαια κοστίζουν και σε χρόνο και σε χρήμα. Η τεχνολογία PEMS είναι πολύ καινούρια τεχνολογία και δεν είναι απολύτως αξιόπιστη ακόμα. Η Επιτροπή Ρουαγιάλ είχε και ως έργο να βελτιώσει, να πάρει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία των συσκευών PEMS. Και αυτό θα γίνει με, το, με τα επόμενα χρόνια. Και οι επενδύσεις μας έχουν αυτό ως στόχο. Έχουμε ε, εργαστήρια, ε, ε, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανεμιστήρες κλπ. που χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλά οι συσκευές PEMS. Οι περισσότερες τεχνικές υπηρεσίες έχουν εργαστήρια γιατί είναι καλύτερο αν θέλει κανείς να είναι εμπειρογνώμονας και ειδικό, ε, αλλά προφανώς χρειάζονται και επενδύσεις. Ehm, Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Τι είδου ε, υπηρεσίες ή παροχές εσείς ε, προσφέρετε στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ή στους κατασκευαστές εξοπλισμών τμήματων αυτοκινήτων. Πέρα από την έγκριση τύπου. Εκτός από την έγκριση τύπου, στο τομέα των δοκιμών, γιατί, όχι, εν γέννη, εν γέννη ρωτάω προτείνουμε στις, στα εργαστήριά μας ε, δυνατότητες δοκιμές, ε, δοκιμών ε, σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα δοκιμών. Υπάρχει μια σειρά νομοθεσιών που πλαισιώνει όλη την αυτοκινητοβιομηχανία και τα πέρα από την νομοθεσία οι κατασκευαστές αλλά και οι κατασκευαστές εξοπλισμών έχουν δικά τους ε, δικές τους απαιτήσεις μπορεί να αφορούν ε, συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε την άνεση, αλλά και δοκιμές κάνουμε που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα προϊόντα. Και πάλι επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο ταχυοταχή, μπορεί να είναι τρακτέρ, φορτηγά, ποδήλατα, οτιδήποτε. Ε, και έπειτα έχουμε κάνει και την ε, έγκριση τύπου συστημάτων διαχείρισης εργοστασίων. Ε, έχουμε πολύ μεγάλο φάσμα δηλαδή εργασιών πέρα από την έγκριση τύπου. Αυτό αντιστοιχεί σε 20% του κύκλου εργασιών μας. Ευχαριστώ. Συνεχίζω ακολουθώντας την τελευταία ερώτηση που υπέβαλε η συνάδελφος. Δηλαδή, χωρίς να είμαι καχύποπτος και χωρίς να θέλω με κανέναν τρόπο να αμφισβητήσω τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό τη εταιρεία σα και των άλλων εθνικών οργανισμών που κάνουν αυτή την εργασία. Εγώ ρωτάω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά. Δηλαδή, ε, ελεγχόμενοι και ελεγκτές ε, έχουν κοινά συμφέροντα. Δεν νομίζετε ότι κάπως θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ των ελεγχόμενων και των ελεγκτών. Κοιτάξτε, η κρίση που μόλις διανύσαμε δεν αφορά τόσο την αξιοπιστία των ε, τεχνικών υπηρεσιών, αλλά τις νομοθεσίες που πλαισιώνουν την πραγματική χρήση ενός οχήματο. Εκεί έγκυται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή περισσότερο από ότι την άλλη πτυχή που εσείς ε, ε, αναφέρεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Κάποιες ερωτήσεις. Στις ε, αναφορές σας ε, αναφέρετε κάποια στοιχεία. Οι νοτιοκοριανικές αρχές βρήκαν μια συσκευή στον Ισανκάσκα. Εσείς έχετε διαπιστώσει ποτέ τέτοιες διατάξεις, τέτοιες συσκευέ σε παρόμοιους ελέγχους. Σήμερα. Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση δεν έχει έρθει ακόμα στο επίπεδο του, της τεχνικής υπηρεσίας. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ακριβώς τι συμβαίνει ανάμεσα στις αρχές Κοιτάξτε, άμα δεν έχετε πληροφορίε τέτοιε, ε, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε στην απάντησή σα. Δεύτερη ερώτηση. Είσαστε η μοναδική τεχνική υπηρεσία στη Γαλλία ε, που ακολουθεί το ιδιωτικό δίκαιο, σωστά. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι, όντω, ναι, καλά κατάλαβα. Ναι, είναι μια ιδιαιτερότητα τη Γαλλία ότι υπάρχει μια μόνο τεχνική υπηρεσία. Ε, εδώ και 45 χρόνια όμω. Μάλιστα. Γιατί αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί, συμβαίνει αυτό στη Γερμανία, τη δική μου τη χώρα. Έχουμε μεγάλο αριθμό τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες είναι και σε μια ανταγωνιστική θέση μεταξύ τους. Συμμετέχει η Γαλλική, το γαλλικό κράτος στην υπηρεσία σας. Όχι καθόλου. Δεν έχει καμία σχέση η εταιρεία μας με το κράτος. Υπάρχει μια ιστορία μακρά που ανανεώνεται καθημερινά. Έπειτα για το πρότυπο δεν νομίζω πως υπάρχει το τέλειο ανάμεσα σε μια διοίκηση και πολλές τεχνικές υπηρεσίες ή μια, μια, ε, ένα διοικητικό μηχανισμό και μια τεχνική υπηρεσία υπάρχουν πολλές πιθανές ε, λύσεις. Ξέρω πως ε, οι αρχές ψάχνονται για να δουν ποιο μοντέλο να ακολουθήσουν στο μέλλον. είναι περίεργο, τουλάχιστον περίεργο, για να το θέσω αυτό ευγενικά, αλλά είναι εντάξει. Έχετε, είστε τυχεροί που δεν έχετε ανταγωνισμό. Μια μικρή παρατηρήση. Από ιστορική άποψη, ε, τα μοντέλα τεχνικού ελέγχου ήταν πολύ συνδεδεμένα με τους κατασκευαστές της χώρας. Και μετά οι τεχνικές υπηρεσίες πέρασαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πελάτες σε κάθε χώρα. Αλλά όντω από ιστορική άποψη οι κατασκευαστέ και ο ρυθμό των κατασκευαστών στη Γερμανία δεν έχει σχέση με τον αριθμό των κατασκευαστών στην Γαλλία. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και την ε, εξήγηση. Η κυρία Γελασέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω επειδή ακριβώς ε, βλέπω ότι μεταξύ σας έχετε και μεταξύ των πελατών σας υπάρχουν και τα φορτηγά όπως η Μπέκο ας πούμε, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε τους εξοπλισμούς για να μπορείτε να ελέγξετε κατά πόσο ο διακόπτης που απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν, έχει, αν σβήνει πριν να μπει στο εργαστήριο που για έλεγχο τον λόγο όχημα. Και έπειτα, Και έπειτα, εσείς μπορείτε να ελέγξετε τα λογισμικά, εσείς δεν έχετε τρόπο, δηλαδή να εντοπίσετε μέσα στα αυτοκίνητα αν ε, ο διακόπτης ήταν στο όνι, ή στο όφο όταν έμπαινε στο εργαστήριο το κάθε όχημα. Excusez-moi, pas bien si votre question est δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Αν η ερώτησή σας δηλαδή αφορά τα φορτηγά ή τα γεωταχή. Φαντάζομαι ότι ακολουθείτε την νομοθεσία γιατί εκεί απαγορεύεται και το επαληθεύεται αν ισχύει όχι. Για τα, γεωταχή, Εφόσον κάνετε αυτή τη δουλειά για τα μεγάλα, για τα φορτηγά, μπορείτε να το κάνετε και για τα, γεωταχή. Το έχετε κάνει σε κάποιες δοκιμές. Έχουμε το υλικό για να κάνουμε δοκιμές για τα φορτηγά σε δικές γέφυρες. για τα χ αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να δούμε, που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να δούμε εάν υπάρχει συσκευή αναστολής, επιμένουμε για την ε, ε, θερμοκρασία, είναι να κάνουμε τις ίδιες δοκιμές σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Τώρα είναι οι δοκιμές ανάμεσα στους 20 και τους 30 βαθμούς, θα μπορούσαμε να τους κάνουμε, κάνουμε τις δοκιμές σε 0 βαθμούς, σε 40 βαθμούς για να δούμε. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξή ότι για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, για εκείνη την νομοθεσία, Περισσότερο μας ρωτούν οι αγοραστές, οι δήμοι ας πούμε για τα λεωφορεία που θέλουν να αγοράσουν. Ανάλογα με τις διάφορες τεχνολογίες και σκέφτονται ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία, μας ρωτούν αν μπορούμε να κάνουμε και δοκιμές ε, εκτός νομοθεσίας, δηλαδή, όπως το RDE, για να δούμε τι γίνεται υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα, λοιπόν, μπορούμε να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε τον πελάτη μας. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γιάλα Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό αν με την ερώτηση. Αν θέλεις. Μπορείς να κάνεις επερώτηση. Όχι, το χρόνο κοιτάω, το χρόνο. Η κυρία Σέντρ χωρίς μικρόφωνο.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 σας ζητούν να εφαρμόσετε τέτοιου είδους δοκιμές, να κάνετε τις ίδιες δοκιμές για τα αυτοκίνητα και τις εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτό, για αυτό το πράγμα έχετε και την αναγνώριση. Για τις είπα, ρωτάτε. Είπα μας αναγνωρίζουν για οτιδήποτε είναι ε, εξοπλισμός. Δηλαδή, φώτα, αερισμός, όχι για το όχημα, όχι. Όχι για τις εκπομπές. Κυρία Σαραντζόβα. Ευχαριστώ πρώτα και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Καταρχά, σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα και για το γεγονό ότι ήλθατε εδώ σήμερα. Όπω ξέρετε, συνεχίζονται οι συζητήσει για το κατά πόσο θα απαγορευτούν τα εργαστηριακά η εργαστηρική έλεγχη στι εγκαταστάσει του κατασκευαστή. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Αναρωτιέμαι, είναι καλή ιδέα αυτή, πιστεύετε, και αν όχι, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ανεξάρτητου ελέγχου ελέγχους ε, στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Και να μας πείτε και δύο λόγια για το τι γίνεται σήμερα που γίνεται πιο πολύ έλεγχη. Απάντηση. Κοιτάξτε, την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε μια αλλαγή στον τρόπο που χορηγούνται οι εγκρίσεις τύπου. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 30-40 χρόνια, οι δοκιμές γίνονταν 100% στα δικά μας εργαστηριά. Με την πάροδο του χρόνου άλλαξε κάπως αυτή η ισορροπία και σήμερα η πλειονότητα των ε, ελέγχων γίνεται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Σήμερα λοιπόν όλες οι δοκιμές που γίνονται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή γίνονται με παρατηρητές, με λεκτές δικούς μας. Δεν ε, εμπιστευόμαστε απλά δηλαδή τα στοιχεία που μας δίνει ο κατασκευαστής. Δεν ε, συμμετέχουμε φυσικά στην διαδικασία κατασκευής του οχήματος. Δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε συνέχεια στον κατασκευαστή. Όταν γίνονται όμως οι δοκιμές στον κατασκευαστή, καταρχάς γίνεται μια επαλήθευση των μέσων, δηλαδή ελέγχουμε όλα τα εργαλεία, όλα τα μέτρα για να δούμε κατά πόσον τα μέσα όντως ανταποκρίνονται στι προδιαγραφέ και λίγο πολύ έχουμε τα ίδια μέσα και στα δικά μας εργαστηρία και άρα έχουμε καλή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη για το τι καταμετράτε και τι μετράτε και πώς. Έχουμε δηλαδή μία αντίληψη ειδικού. Ευχαριστώ. Κυρία Γκροστέτ, σας ευχαριστώ. Μας είπατε πριν από λίγο ότι θέλετε να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου. Αυτό τι σημαίνει, ότι πιστεύετε ότι μια έγκριση τύπου χορηγείται πιο εύκολα σε κάποιο κράτος μέλος από ό,τι σε άλλα και ως τεχνική υπηρεσία, ως τεχνικές υπηρεσίες γίνεται, κάνετε ανταλλαγές ε, βέλτιστων πρακτικό. Απάντηση, κοιτάξτε, οι ερμηνείε μπορεί να είναι διαφορετικές. Ναι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, το έχουμε βιώσει άλλωστε. Σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές τώρα. Όπως σας είπα, εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχουμε στην κατάρτιση της νομοθεσίας και στην, ομο... στην ομάδα αυτή έχουμε τους ομολόγους μας από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία και άλλα άτομα της τεχνικής υπηρεσίας και όντω. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε ως τεχνικές υπηρεσίες μια κοινή ενιαία θέση για το πώς θα ερμηνευτεί το χύψη στοιχείο υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών για να υπάρχει καλύτερο συντονισμό σε ό,τι αφορά την έκδοση τύπου. Να συνεχίσω λοιπόν γρήγορα γρήγορα. Τι οχήματα χρησιμοποιούνται για την διενέργεια των έλεγχων που απαιτούνται. Και μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι δεν πρόκειται για βελτιστοποιημένα οχήματα τα οποία είναι πειραγμένα τελευταία στιγμή για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στους ελέγχους. Είστε βέβαιοι γι' αυτό. Απάντηση. Ακόμα και αν υπήρχαν αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου, θεωρώ ότι δεν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτό, γιατί αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι ότι ένα συγκεκριμένο όχημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μας διαβιβάζει ο κατασκευαστής είναι πιο πολύ μας απασχολεί το θέμα και το σκέλος της ε, κατασκευής. Η έγκριση τύπου για ένα όχημα θα χορηγηθεί σε τελική ανάλυση, αν όχι σήμερα, αύριο. Αλλά αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι κατά πόσον αυτό που εγκρίθηκε τελικά είναι αυτό που παράγεται, αυτό που κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ κυρία Πουνεφά. Σας ευχαριστώ. Κάπου έχασα την ερώτησή μου. Τη βρήκα. Δύο ερωτήσεις έχω και πρέπει να βιαστώ κιόλας. Πρώτη. Είπατε ότι για να ανταποκριθείτε στις τα αιτήματα της Επιτροπής Ρουαγιάλ ε, αναπτύξατε το σύστημα PEMS. Το σύστημα PEMS φορητού συστήματος μέτρησης εκπομπών. Πόσο καιρό το έχετε? Πόσο καιρό το χρησιμοποιείτε? Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε τη σχετική ρύθμιση RDE χρησιμοποίησαμε τα PEMS, αλλά δεν ήταν ε, τα, της τελικής μορφής PEMS. Ε. Ήταν κάποια αρχικά φορητά τέτοια συστήματα μέτρησης εκπομπών. Όπως είπε και ο κ. Μπενουά, όταν κάναμε τους ελέγχους για την Επιτροπή Ρουαγιά, ε, παραβλέψαμε και αφήσαμε κατά μέρον αρκετά στοιχεία για, για τα αποτελέσματα. Τα χρησιμοποιούσαμε λοιπόν για να αναπτύξουμε τη μέθοδο, γιατί συμμετείχαμε στη διαδικασία κατάρτισης μια μεθόδου, αλλά επισήμως στα πλαίσια της Επιτροπής έγιναν αυτά. Μάλιστα. Και στις απαντήσεις σας προς τους συναδέλφους είπατε σε πολλές περιπτώσεις ότι ακολουθείτε απόρριτα την νομοθεσία και συμφωνούμε μαζί σας. Αυτή η ρύθμιση γίνεται λοιπόν βάσει της ε, τιμές ε, εκπομπών οξυδίου του άνθρακα και οξυδίου του αζωτού. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Και είναι σημαντικό να ακολουθείτε και η νομοθεσία, για παράδειγμα, για την ασφάλεια των οχημάτων. Για τα φρένα, για παράδειγμα. Υπάρχει μια νομοθεσία για την έγκριση τύπου. Υπάρχουν λοιπόν για τέτοια θέματα ασφαλείας ε, ε, τέτοιες διατάξεις. Υπάρχει κάποια διαφορά σε ό,τι αφορά αυτή τη διατάξη για το περιβάλλον ή σε ό,τι αφορά τις διατάξεις ασφαλείας. Θέλω δηλαδή να μου πείτε αν μόνο για θέματα ρήπανση επιτρέπεται η υπέρβαση δύο και τρεις φορές των ορίων που προβλέπονται για τις εκπομπές και είναι πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι σε σχέση τα φρένα για παράδειγμα. Κοιτάξτε. Είναι περιπλοκή η απάντηση, αλλά προφανώς και για θέματα ασφάλειας και για θέματα περιβάλλοντος θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές. Αλλά μας είπαν προηγουμένως ότι οι κατασκευαστές χρειάζονται χρόνο για να ανταποκριθούν στα επίπεδα που προβλέπονται, αλλά ε, υπερβαίνονται κατά δύο φορές ενδεχομένως τα όρια Αναρωτιέμαι, την ίδια ευελιξία, την ίδια ανοχή δείχνουμε και για τα πρότυπα που προβλέπονται για θέματα ασφαλείας όπως είναι τα συστήματα πέντησης. Κοιτάξτε, για τα θέματα ασφάλειας υπάρχει το Euro Cup, μια προδιαγραφή η οποία ξεπερνάει τα θέματα κανονιστικής ρύθμισης. Αυτό χρησιμοποιείται από όλου του κατασκευαστέ στην Ευρώπη. Και η ρύθμιση προέρχεται από το ONCAP. Και να σα πω δύο λόγια. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όπως υπάρχει στα θέματα ασφάλειας για τα PEMS. Η τεχνολογία ε, φυσικά χρειάζεται και κάποιο χρόνο να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όπως αυτό που υπάρχει σε θέματα ασφάλειας. Η κυρία, ο κύριος Γκίζικε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπενουά, κυρία λόπε, σας ευχαριστούμε που ήλθατε εδώ σήμερα για να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά και θα ήθελα να επανέλθουμε στο θέμα της χειραγώγηση του λογισμικού. Κύριε Μπενουά, είπατε ότι δυστυχώς εδώ σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και τον εντοπισμό τη απάντησης δεν έχουν σημειωθεί εξελίξει 380 ε, μηχανικοί είναι στην ε, επιχειρή σας. Πόσοι είναι ειδικοί σε θέματα λογισμικού μεταξύ αυτών. Πολύ λίγοι. Δεν είναι ένας ε, τομέας ε, στον οποίο η νομοθεσία απαιτεί από εμά να έχουμε πολύ προσωπικό και να είμαστε ισχυροί δεν έχουμε χτίσει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα. Η Επιτροπή Ρουαγιάλ ε, μάλιστα ανέθεσε στο ε, εργαστήριο Λίσπεν το θέμα της, ε, του ελέγχου του λογισμικού και όχι σε εμάς. Ακριβώς διότι εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ ειδικευμένοι. Αν κάποια στιγμή η νομοθεσία μας υποχρεώσει να κάνουμε περισσότερους ελέγχους λογισμικού, ασφαλώς ε, θα εμβαθύνουμε. Πάντως είναι πολύ περίπλοκο. Επιτροπές που συστάθηκαν σε διάφορες ε, χώρες προσπάθησαν ε, να εντοπίσουν λογισμικά έτσι ύποπτα, αλλά δεν έχουν πετύχει από όσο ξέρω. Γιατί, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο να εντοπιστεί αυτό το παράτυπο λογισμικό. Σας ευχαριστώ για την απάντηση αυτή η οποία δεν ε, είναι και βασίζεται και στο μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε ενδεχομένω γι' αυτό ακόμα και δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι ειδικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά συστήματα με τις εκπομπών, στην Επιτροπή ε, ακούσαμε διάφορους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας λένε ότι υπάρχει ακρίβεια 10 20%. Εσείς μας λέτε ότι η ακρίβεια απέχει κατά πολύ από το 100%. Πώς αξιολογείτε λοιπόν τις μετρήσεις των ΠΕΜΣ. Είναι αξιόπιστες αυτές οι διαφορετές ε, συσκευές μέτρησης εκπομπών. Καταρχήν έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, η αξιοπιστία του ίδιου του οργάνου η οποία βελτιώνεται σιγά σιγά ε, από τους κατασκευαστές τους. Ε, στην Επιτροπή Ρουαγιάλ ε, πολλές φορές χρειάστηκε να επαναλάβουμε δοκιμές γιατί το αποτέλεσμα που είχαμε πάρει με το, τη συσκευή πέμψη δεν ήταν καλό γιατί δεν είχε λειτουργήσει καλά. Μετά την επόμενη φορά λειτουργεί σωστά. Ε, 20% έξω πέφτει. Ε, δηλαδή έχει ακρίβεια συμπλήν 20% το όργανο αυτό. Οπότε ε, αυτή τη στιγμή τώρα θα βελτιωθεί. Αλλά ποτέ δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα ακρίβειας εργαστηρίου. Ε, Απ' την άλλη μεριά, η, η αξιοπιστία των ίδιων των συσκευών σε ό,τι αφορά το αν δουλεύουν ή όχι σωστά ε, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Thank you very much. Um, maybe Μια τελευταία ερώτηση νομίζω ότι έχω. Δεν καταλαβαίνω πια τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται με εγκριστή που η αρχή που σα ζητάει εσά που είστε τέχνη από εσά που είστε τεχνική υπηρεσία, να κάνετε τι δοκιμέ, οι οποίε περιγράφονται λεπτομερώ. ε, και αν περάσει το αυτοκίνητο τι δοκιμέ αυτέ, εγκρίνεται και βγαίνει στην κυκλοφορία. Όμω, οι αρχέ εγκριστή τύπου πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι, συμμορφώνονται σε κανονική χρήση, άρθρο 5 του κανονισμού για την ποιότητα του αέρος. Οπότε σε κανονική χρήση θα πρέπει οι εκπομπές να είναι χαμηλότερες των ορίων ε, και, οι, και απαγορεύονται οι διατάξεις αναστολή. Ποιος είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή αυτού του κομματιού της νομοθεσίας. Ότι δηλαδή τα αυτοκίνητα συμμορφώνονται με αυτό το κομμάτι τη νομοθεσία. Ποιο το ελέγχει. Ε, είπαμε, εμείς ασχολούμαστε με την συμμόρφωση παραγωγής, με την έγκριση τύπου και ε, αυτά είναι που μας υποχρεώνει η νομοθεσία. Ε, δεν σας αρέσει αυτό θα σας πω, αλλά το άλλο κομμάτι, την χρήση την χρήση κανονική λειτουργία, δεν έχει, δεν έχει αναπτυχθεί αυτό και η RDE, αυτή η μέθοδος μέτρησης των εκπομπών στο δρόμο, ε, αποσκοπεί ακριβώς προς αυτό. Να δούμε τι γίνεται μετά. Ε, με αυτή τη μέθοδο πράγματι περνάμε σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Ε, καταλαβαίνω ότι λέτε δεν, είναι τμήμα του, δεν ήταν μέχρι τώρα τμήμα της έγκρισης τύπου, το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, αλλά ο νομοθέτης πρέπει να κάνει και κάτι παραπάνω από έγκριση τύπου, γιατί ε, άπαξ και το αυτοκίνητο βγει στους δρόμους, κανείς δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί οι κανόνες είναι, υπάρχουν. Λένε, απαγορεύονται διατάξεις αναστολής. Ποιος είναι υπεύθυνο αρμόδιος έτσι ώστε να τηρείται αυτό το κομμάτι τη νομοθεσία. Απάντηση. Οι αρμόδιε αρχές σε θέματα ε, τύπου. Οι εθνικές αρχές εγκριστήπου. Έχουμε εδώ ένα, ένα εκπρόσωπο τέτοια ε, αρχή, οπότε θα τον ρωτήσουμε πώς κάνει τη δουλειά του. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Όχι. Εντάξει. Ε, τελειώσαμε με την ε, ακρόση αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Ίσως υποβληθούν και γραπτές ερωτήσεις. Ε, η προθεσμία για την υποβολή τέτοιων γραπτών ερωτήσεων είναι 17 Οκτωβρίου.

colleagues, uh, let's proceed for the last hearing of... Uh, Περνάμε στην τελευταία μας ακρόαση για σήμερα. Ξεκινήσαμε ήδη από χτες το απόγευμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι η μεγάλη τιμή μα που προσκαλούμε και υποδεχόμαστε εδώ πέρα τον κύριο Ρέιντερ και τον κύριο Βάλκ, ε, ε, του Ολλανδού εκπροσώπου του RDV. Χαίρομαι που δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μας. Θα δίνει το λόγο και μετά θα πάρουν το λόγο και οι βουλευτέ για να θέσουν ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί βουλευτέ, και κύριοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Όταν διάβασα το άρθρο για την υπόθεση Volkswagen το Σεπτέμβριο 2015 στον τύπο, κατάλαβα ότι τα μέσα ενημερωσής δεν ασχολιόντουσαν μόνο για τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και την πραγματική ε, κατανάλωση σε σχέση με το εργαστήριο, αλλά και για τις ε, εκπομπές οξυδίου του, οξυδίων του αζότου από τα αυτοκίνητα diesel. Τότε όμως δεν μπορούσα να προβλέψω πόσο σημαντικός θα ήταν ο αντίκτυπος για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. διότι ε, έδωσε τη, μια όθηση στην ανάπτυξη του δεύτερου πακέτου της, ε, ε το, της διαδικασίας RDE που βρισκόταν στο, στη δεύτερη φάση της ε, και περιμέναμε τις προτάσεις κομισιών. Ε, η Επιτροπή σας μου δίνει την ευκαιρία να σας ενημερώσω για το πώς, έχει συμβάλει, πώς έχουν συμβάλει κάτω χώρε και η RDW στην βελτίωση των κανόνων ιδιαίτερα για τις διαδικασίες μέτρησης ε, κομπών. Ε, Ονομάζουμε Rangers Αντρέ ε, Ρέιντερς, είμαι σύμβουλος εκπομπών και, και καυσίμων οχημάτων στην ε, ε, υπηρεσία οχημάτων της, ε, των κατοχωρών. Είναι μια, ένας φορέας που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υποδομών, απασχολεί περίπου 1.400 άτομα και έχει ως αποστολή ε, η αποστολή της αφορά την, ε, την έγκριση τύπου ε, οχημάτων και εξαρτημάτων τους, ε, παροχή πληροφοριών, ε, έκδοση εγγράφων όπως οδειών και κλπ. Δεν είμαστε λοιπόν μόνο ένας φορέας έγκσης τύπου. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Η RDW συμμετέχει σε διάφορα διεθνή φόρα στον Οργανισμό Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όπου ε, τυχάνουν επεξεργασία νομοθετικά κείμενα που αφορούν τα οχήματα. Έχουμε ένα ε, τμήμα μάλιστα ε, από οκτώ εμπειρογνώμονες ε, που ασχολούνται ακριβώς με αυτή μας την συνεισφορά σε διάφορους τομείς. Εγώ είμαι ο εμπειρογνώμονας για το θέμα των εκπομπών οχημάτων. Είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΟΗΕ για το θέμα της εναρμόνισης των κανονισμών ε, οχημάτων στη Γενέβη. Επίσης, στις Βρυξέλλες δρώ ως εθνικός τεχνικός εμπειρογνώμονας για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Μεταφορών και Υποδομών, συγγνώμη. Και μάλιστα συμμετέχω και σε διάφορες ομάδες εργασίας μεταξύ αυτών και η Τεχνική Επιτροπή ε, ε, Οχημάτων τη CMV. Εξετάζοντα τον ε, κανονισμό εκπομπών ε, Euro 5 και Euro 6 στην Ευρώπη, ε, ο οποίο υιοθετήθηκε από... υιοθετείται με συναπόφαση ε, 752 του 07 συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις, τις γενικές διατάξεις, όχι ειδικέ διατάξεις, για, τα καυσαέρια, για τις εκπομπές αυτοκινήτων. Τα εφαρμοστικά μέτρα περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που υιοθετούνται μέσω της ε, τροπολογίας. Είναι ο εφαρμοστικός κανονισμός 692 του 2008. Στην διαδικασία έγκρισης τύπου η τεχνική υπηρεσία ελέγχει ε, την συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών και μετρά τις, ε, με τις εκπομπές διοξυδίου του ε, άνθρακα μέσω του NEDC. Κανένα άλλο, ε, καμία άλλη δοκιμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης. Προκειμένου να αποφύγουμε διαφορές μεταξύ των μετρήσεων που κάνουν διάφορες τεχνικές υπηρεσίε. Όπως γνωρίζετε, αυτός ο κύκλος δοκιμών έχει ηλικία άνω των 20 ετών και δεν είναι προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα. Για το διοξείδιο του ανθρακά το 2017 αυτός ο κύκλος θα αντικατασταθεί από ένα καινούριο. Είναι ε, η διαδικασία WLTP. Η ανάπτυξη αυτού του νέου κύκλου δοκιμών γίνεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Εθνών η, στο πλαίσιο, στο πλαίσιο μιας εργασίας που ξεκίνησε ήδη από το 2010. Η RTW προσωπούσε τις ε, κάτω χώρες από την αρχή ε, έτσι ώστε η WLTP να μπορέσει να μεταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το 2006 όμως, πιο πριν, κατά τη διάρκεια της ε, επεξεργασίας των βασικών αρχών για το Euro 5 και Euro 6, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη είχε προβλέψει ότι οι δοκιμές NEDC δεν θα είναι επαρκείς ούτε και για τα οξύδια του αζότου και άλλους ρήπους. Αυτό από το 2006. Η Κομισιόν ε, είχε σκεφτεί τη χρήση των PEMS έτσι ώστε τα οχήματα να δοκιμάζονται στο δρόμο. Με το άρθρο 14.3 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να αναπτύξει, να επεξεργαστεί τέτοια νομοθεσία μέσω της ετροπολογίας. Η επεξεργασία αυτή ξεκίνησε το 2011, 4,5 χρόνια λέει, περίπου πριν την υπόθεση Volkswagen. Εγώ προσωπικά είχα ε, συμμετάσχει από την αρχή έτσι ώστε να εξασφαλίσω ότι θα εκφράσει σωστά η άποψη των κατοχωρών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ε, αρκετές ολλανδικές προτάσεις έγιναν δεκτές ε, στο πλαίσιο των τεχνικών διατάξεων του πρώτου και του δεύτερου πακέτου RDE που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το Μάιο το πρώτο και τον Οκτώβριο του 2015 το δεύτερο. Όμως το αποτέλεσμα του δεύτερου πακέτου RD από τις τελευταίες διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Επιτροπή μας ε, δεν αντικατοπίζει ακριβώς τις Ολλανδικές θέσεις. Για παράδειγμα, η ημερομηνία θέση εφαρμογή ε, που, που αναβλήθηκε κατά ένα έτος και η αύξηση του συντελεστή συμμόρφωσης 1,6 που αυξήθηκε στο 2,1 ε, δεν μας ικανοποιούσε και αυτό λόγο ψηφίσαμε κατά το αποτελέσμα στο τελικό αποτέλεσμα της όλα αυτά, θέλω να καταστήσω σαφές ότι ε, μας ικανοποιεί που έχουμε δύο πλέον εφαρμοστικούς κανονισμούς για την διαδικασία RD. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τελευταία φάση του τρίτου πακέτου RDE δηλαδή, θα ολοκληρωθεί στην TCMB σύντομα. Και εκεί έχουμε ζητήσει ε, βελτιώσεις και έχουν συμπεριληφθεί. Ένα σημαντικό τμήμα όμως αυτής της νομοθεσίας RD θα είναι το τέταρτο πακέτο RD ε, που δίνει την δυνατότητα πρόσθετων δοκιμών RDE από ανεξάρτητους φορείς σε δημόσιους δρόμους. Αυτό ε, μπορεί να ειδωθεί ως τμήμα της εποπτείας αγοράς. Στο πλαίσιο του καινούργιου κανονισμού έγκρισης και εποπτείας αγοράς. Η RDW είναι, ε, συμμετείχε στην διαδικασία αυτή, εκφράζοντα τι ε, απόψει των χώρων, Δεν είμαι εμπειρογνώμονα, δεν είμαι ειδικό για αυτό το θέμα, οπότε μπορώ να σα ενημερώσω μόνο γενικά. Οι κάτω στηρίζουν τι προθέσει αυτή τη πρόταση. Είμαστε σίγουροι ότι στόχο είναι η βελτίωση του συστήματο έγκριση και η βελτίωση της, ε, του επίπεδου εποπτείας αγοράς είμαστε επικριτικοί σε σχέση με ορισμένε από τι λύσει που επιλέχθηκαν και έχουμε προτείνει άλλε λύσει που πιστεύουμε ότι είναι πιο αποτελεσματικέ και πιο ρεαλιστικέ και εξασφαλίζουν ταυτόχρονα το ίδιο επίπεδο βελτίωση. Μετά την υπόθεση Volkswagen έχει δημιουργηθεί μια καινούργια πραγματικότητα. Και το Εθνικό μα Κοινοβούλιο έχει δείξει ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα υποβλήθηκαν τρεις ερωτήσεις και τρεις προτάσεις ψηφισμάτων. Αυτό ενθαρρύνει, μας ενθαρρύνει στη θέση μας. Ενισχύει τη θέση μας. Ε, και θέλουμε να βελτιωθεί το επίπεδο εποπτείας. Τελειώντας να επιβεβαιώσω ότι η RDW θα συνεχίσει να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ε, ε, επεξεργασία της βέλτιστης ε, της νομοθεσίας και θα συμμετάσχουμε ε, στην την άποψή μας στην συζήτηση όλων των κανονισμών για τη διαδικασία RD. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Uh, σας ευχαριστώ και θα δώσουμε τον λόγο κατευθείαν στον εισηγητή μας, τον κύριο Χερμπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και ιδιαίτερω τον κύριο Ρέντερς και τον κύριο Βάλτη για την παρουσία τους εδώ για τη... τα σχόλια τους, τα εισαγωγικά του σχόλια. Μία ερωτήση. σε ό,τι αφορά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι τόσο επισταμένος εδώ και μια μισή μέρα. Λέτε ότι στον κανονισμό δεν υπάρχει οποιαδήποτε προδιαγραφή για την ε, ανείχνευση απαγορευμένων διδάξεων αναστολή. Αυτό είναι ο λόγο που αναφέρεται για τον οποίο δεν γίνονται ελεγχοί. Αυτό λοιπόν αποτελεί τον φαύλο κύκλο αν θέλετε γιατί δεν υπάρχουν λοιπόν τεστ για τον εντοπισμό διδάξεων αναστολή. Άρα δεν θα βρίσκουμε. Για τον νομοθέτη και για τις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Ιδιαίτερα επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι διατάξεις αποστολής εδώ και χρόνια, αναστολής εδώ και χρόνια. Έχουμε καλές επαφές με τον φορέα που εντοπίζει τις πρακτικές αυτές εδώ και καιρό στην Ευρώπη. Ερωτώ λοιπόν, με τι τρόπο προσπαθήσατε αυτό το cycling beating, τις διατάξεις αναστολής να τις εντοπίζετε, γιατί θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τμήμα των αρμοδιοτήτων των Ολλανδικών αρχών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή που μας θέτετε. ορισμός και η αξιολόγηση μιας διαταξής αναστολής είναι πάρα πολύ δύσκολος και αυτό προκύπτει διαρκώς ε, και στη συζήτηση που έγινε σήμερα και στις προηγούμενες ακροάσεις. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να α, θεωρήσει ο κατασκευαστής ως ε, μέθοδο πειράγματος, χειραγώγησης. Και αυτό είναι καταριστικό στις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναζητήσει κανείς τρόπους ε, πειράγματος. Από πού να ξεκινήσουμε πώς θα μπορούσε να έχει εντάξει ένα τέτοιο σύστημα ο κατασκευαστής σε ένα όχημα. Το να αναζητήσει λοιπόν κανείς κάτι το οποίο δεν ξέρει τι υπάρχει είναι πάρα πολύ δύσκολο, ψήλο στα χειρά. Και γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή στην νομοθεσία Euro 5 και στην διαδικασία επιτροπολογίας σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμπληρωματική μέθοδος ελέγχου πέρα από το RDC e το NDC e συγγνώμη, στα εργαστηρία. Και αυτό ήταν ένας από τους στόχους της σύστασης του, του ελέγχου RDE για να μειωθεί ο αντίκτυπος των διατάξεων αναστολής. Το κατανοώ αυτό για το μέλλον. Δηλαδή από το 2007 όμως και μετά Έχουμε απλά σηκώσει τα χέρια ψηλά και λέμε ότι οι διτάξεις αναστολής δεν θα εντοπίζονται μέχρι ότου ε, περάσουν οι, τα τεστ πραγματικών εκπομπών. Δέκα χρόνια δηλαδή. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δεν είναι καθήκον των Ολλανδικών αρχών του νομοθέτη και μάλλον της αρχής επιβολής της ε, νομοθεσίας να διασφαλίσουν ότι θα εντοπιστούν αυτές οι διατάξεις μέσω πιο πολύ σύνθετων τεστ, για παράδειγμα. Δεν λάβατε ποτέ σχετική εντολή. Δεν το κάνατε αυτό. Αυτό ακριβώς που λέτε, το τελευταίο. Όλοι ξέρουμε και κατέστησα θέση ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των τεστ στα εργαστήρια και στον ε, δοκιμών στον δρόμο. Αυτό που διαπιστώσαμε με τις φορτές, ε, με τα φορτές συστήματα μέτρησης εκπομπών. Και όλα αυτά προέκυψαν το 2010, τον Νοέμβριο, σε μια σχετική μερίδα, η οποία διοργανώθηκε εδώ στις Φρυξέλλες. Καταδείχθηκε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δοκιμών και του, των δοκιμών στον δρόμο. Και είπαμε ότι θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το χάσμα γιατί πολύ απλά δεν συνάδει με τους στόχους της ε, νομοθεσίας για τις εκπομπές. Άρα, όλοι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην διενέργεια τέτοιων ελέγχων που θα αποτύπωναν τα πραγματικά αποτελέσματα. Η αναζητήση των διατάξεων αναστολή δεν αποτέλεσε κατεξοχήν και κάθε αυτό στόχο. Υπήρχε εμπιστοσύνη και το εννοώ, το εννοώ. Υπήρχε εμπιστοσύνη ότι ο κατασκευαστή δεν θα έκανε σκόπιμα κάποια χειραγώγηση. Μάλιστα, άρα τώρα θα πρέπει να είστε λογικά εξοργισμένοι, γιατί αυτή η εμπιστοσύνη έχει καταπατηθεί κατάφορα. Όχι μόνο στη Volkswagen, αλλά και στη Fiat, αλλά και σε άλλου. Φαντάζομαι λοιπόν ότι το μετανιώνετε πικρά που εννέα χρόνια τώρα δεν κάνετε πιο αυστηρούς ελέγχου. Σα ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο ως μοναδική αρχή σε όλη την Ευρώπη να ξεκινήσουμε μία έρευνα φέροντας ότι κάτι πάει στραβά. Νομίζω ότι στην Ευρώπη υπάρχει ενιαία αγορά, συνεργαζόμαστε με όλα τα εντρήματα και αν από πλευράς πολιτικής και από τις έρευνες TNO στην Ολλανδία και στην Εθνική Βουλή προκύψει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις διαφορές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τους εργαστηριακούς και στον δρόμο. Δεν ήταν καν στην ημέρια διάταξη το θέμα. Άρα, αυτό καταλαβαίνετε τι κάνει στην ε, ανάγκη αναζητήσει κάτι που δεν ξέραμε καν τι υπάρχει. Ο κύριος Κίσεκε. Ευχαριστούμε Κύριε Ρέινερς, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα αυτό και πολύ τεχνικό. Ναι, δεν μιλάω Ολλανδικά. Θα, θα μιλούσα Ολλανδικά μου μπορούσα, αλλά θα μιλήσω Γερμανικά και θα χρειάζεται την πολύ. Φοβάμαι. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά, όχι μόνο τα τεχνικά, αλλά και τα θέματα αρμοδιοτήτων και κατανομής των αρμοδιοτήτων στα κρατημέλη. Είσαστε σύμβουλος όντως ανεξάρτητος ή είστε δημόσιος υπάλληλος. Αυτό είναι μια πρώτη ερώτηση για το ποιος είστε ακριβώς. Ποιος είναι αυτός που μας απευθύνει το λόγο. Είμαι ο Άντρι Ρέιντερς. Αυτό πρώτο και καλύτερο. Και εργάζομαι στην RDV. Στην υπηρεσία Που έχει την έντολη και την αρμοδιότητα από Ολλανδικής πλευράς να κάνει τεχνικούς ελέγχους σε συντονισμό με το Εθνικό Υπουργείο αλλά εκπροσωπούμε και την Ολλανδία στα διεθνή φορά. Παρά το γεγονός ότι είμαι υπάλληλο της RDW. Εκπληρώνουμε λοιπόν ε, δημόσια καθήκοντα, απαντάω έτσι στα ερωτήματά σας. Ναι, είμαι δημόσιος υπάλληλο. Ναι, αυτή ήταν η σωστή και πιο ακριβής απάντηση, ότι είστε δημόσιος υπάλληλος. Αλλά θα σας ε, εμπιστευόμουν ακόμα και αν ήσασταν απλός ομπειρογνώμονα. Δεν ήταν αυτό που με απασχολούσε. Σήμερα και χθε ακούσαμε συναδέλφου σας ε, εμπειρογνώμονες από το Λουξεμβούργο, την Ιταλία και αναφέρθηκε η χρήση θερμικών παραθύρων, διατάξεων αναστολής που αυτόματα θέτει εκτός λειτουργίας το σύστημα να κυκλοφορήσει μετά από 22 λεπτά. Και αναφέρθηκε από το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι και νόμιμο. Με διαφορετικό λοιπόν τρόπο ερμηνεύεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πώς κρίνετε εσείς το θέμα αυτό, για παράδειγμα, του θερμικού παραθύρου των διατάξεων αναστολή που αναπροερχοποιούνται μετά από 22 λεπτά από ενεργοποιούν το σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαέριων. Πιστεύετε ότι αυτά είναι σύνομο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Μετά από όλε τι έρευνε που έχουν γίνει μετά το σκάνδαλο της Volkswagen από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο όλες αυτές οι χώρες ξεκίνησαν έρευνες. Αυτό που προκύπτει από τις έρευνες είναι ότι σαφώς υπάρχουν ε, πολλές ε, περίεργες μορφές, περίεργες μορφές ελέγχου των εκπομπών. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει τώρα είναι κατά πόσον όλες αυτές οι στρατηγικές είναι αποδεκτές ή όχι. Αν πρόκειται για πραγματική διατάξη αναστολής ή όχι και κατά πόσον ο κατασκευαστής μπορεί να καταδείξει ότι αυτή η διάταξη έχει σκοπό την προστασία του κινητήρα ή αν η τεχνολογία αυτή είναι ανεπαρκής για να ρυθμίσει μέσα στο τρόπο την εκπομπή καυσαέριων. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που ανακύπτουν και έρχονται στην επιφάνεια. Το θέμα λοιπόν είναι να καθοριστεί και πάλι μια κοινή τοποθέτηση στην Ευρώπη για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικός κρίκος για την διεξαγωγή των συζητήσεων αυτών με τις διάφορες αρχές έγκρισης τύπου που έκαναν τις σχετικές έρευνες. Και εδώ αναζητούμε μία αξιολόγηση για το ποιες ε, διατάξεις ε, χρησιμοποιήθηκαν για χρήσεις οι οποίες δεν είναι αποδεκτές και θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως παράνομες διατάξεις αναστολής. Ελπίζω έτσι να απαντώ στην ερώτησή σας. Oh, Συνεχίζω πάνω στο θέμα της, ε, των, των διατάξεων αναστολής και την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 8. Εδώ μιλάτε για κάτι το οποίο προκάλεσε τον ενδιαφέρον μου, φαντάζομαι πως δεν είμαι η μόνη. Ε, πρόκειται για τις κατευθυντήριες γραμμές για το DRC Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εντοπισμό ε, διατάξεων αναστολής. Δεύτερη γραμμή στην απάντησή σας. Ποια ερώτηση είπατε, σελίδα 6, ερώτηση 8, είναι η δεύτερη σειρά της απάντησής σας. Λέει, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τις κατευθύνσεις γραμμές για να κάνουμε τις πλέον δοκιμές. Ναι, σαφές. Ε, συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να ψάξω πού βρισκόμασταν ακριβώς. Πρόκειται για τη συνέχιση της ε, απάντησης την οποία έδωσα πριν από λίγο. Έγιναν διάφορες ε, έρευνες, δημοσιεύτηκαν και τα αποτελέσματα και τα απορίσματα της έρευνας. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξή. Στην Ευρώπη θα πρέπει να δρούμε με έναν ενιαίο τρόπο και να καθορίζουμε τα επόμενα βήματα μας. Τα επόμενα βήματα μπορούν να καθοριστούν μόνο αν τα αποφασίσουμε από κοινού. Έτσι δουλεύουμε εδώ στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει ότι μεταξύ Γερμανίας, Αγγλίας και όλων των άλλων που έκαναν σχετικές έρευνες θα πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και τονίσαμε, το ζητήσαμε κιόλα να λάβουμε κατευθυντέρες γραμμές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μας το υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Συμβουλίο Μεταφορών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ε, χρησιμοποιήσατε, ακολουθήσατε αυτή τη μεθοδολογία του GRC. Αυτό λέτε στην απάντησή σας, το χρησιμοποίησατε. We used. Είχατε τα πρώτα αποτελέσματα, μπορούν και αυτά να δημοσιευθούν, να δημοσιοποιηθούν, μπορείτε να μας τα δώσετε αναλυτικά. Ναι, το JRC βοήθησε για να περιγράψουμε το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο οι έλεγχοι. Πιο γρήγορα, πιο αργά. Με άλλες ταχύτητες. Οποιασδήποτε άλλες μορφές ε, για τον εντοπισμό περίεργων συμπεριφορών. Το κάναμε λοιπόν αυτό ως RDW. Να σας πω ότι τότε που ξεσπάσε το σκάνδαλο της ε, Volkswagen, το RDV, έθεσε κατευθείαν το ερώτημα. Ήταν πραγματικά η μοναδική εταιρεία, η Volkswagen. Νομίζω ότι όλοι αναρωτήθηκαν γι' αυτό. Και εμεί ε, χορηγήσαμε έγκρισης τύπους. Ναι, συγγνώμη, η συγκεκριμένη ερώτηση όμως που σας ε, απέθυνα είναι κατά πόσον το χρησιμοποιήσατε αυτό σε κάποιο όχημα και κατά πόσον ανακλήθηκε έγκριση τύπου από όχημα γιατί είχε χρησιμοποιήσει διατάξη αναστολή. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη ερώτηση που έθεσα. Όχι. Θέσαμε μόνο ερωτήσεις προς τους κατασκευαστές για την ε, χρήση διατάξεων αναστολή όπως αυτές που χρησιμοποίησε η Volkswagen. Όλοι απάντησαν αρνητικά και έτσι συνεχίσαμε με το οργανωμένο πρόγραμμα όπως αυτό που προβλεπόταν από το ERC. Ε, ελέγξαμε λοιπόν 30 οχήματα. Η έκθεση σχετική ολοκληρώνεται όπου να είναι. Θα αποσταλεί μέσα στο μήνα στην Εθνική Βουλή. Και στη συνέχεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Και ενώπιν της Επιτροπής μας μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον κάποιο όχημα είχε χρησιμοποιήσει διάταξη αναστολή σε ό,τι αφορά την έκθεση την οποία θα δημοσιεύσετε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβώ σε σχετικές δηλώσεις γιατί θα πρέπει πρώτα να κατατεθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο η έκθεση αυτή και μόνο τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα πορίσματα. Και την επόμενη μέρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσθέτει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Γερμπράντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάτι συγκεκριμένο. Έχετε κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη στην οποία θα υποβληθεί στην Εθνική Βουλή η έκθεση. Όχι, δεν έχω την ακριβή ημερομηνία. Μέσα στο μήνα όμω, στο τέλη του μήνα, μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ, γιατί κατά το παρελθόν είχαμε ακούσει ότι θα γινόταν αυτό και το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, για πείτε μα, τι θα κάνουμε με τα οχήματα τα οποία αποδεδειγμένα δεν συμμορφούνται με την ε, νομοθεσία και έχουν λάβει παρόλα αυτά έγκριση τύπου. Το RDV ε, μπλέκεται με το Opel Σαββίρα. Διάφορες έρευνες κατέδειξαν ότι είναι πολλαπλάσεις οι εκπομπές του από τις επιτρεπόμενες, άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και το RDV έδωσε την οριστική έγκριση τύπου και αληθεύει ότι το RDB μπορεί μάλλον να ανακαλέσει τέτοια έγκριση τύπου εφόσον χρειαστεί. Το RDV έδωσε μόνο τη γενική έγκριση τύπου. Σε ό,τι αφορά α, την έγκριση για τις εκπομπές, αυτή χορηγήθηκε από το ΚΑΜΠΕΑ και η οποία έκανε έρευνα βάσει του Opel Zafira. Συμμετείχε και το RTV στις μελέτες αυτές, τις έρευνες αυτές, αλλά μπορούμε να δράσουμε και να ενεργήσουμε μόνο αυτή τη στιγμή. Λάβουμε πληροφορίες περαιτέρω από την ΚΑΜΠΕΑ για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν γιατί εδώ μιλάμε για την έγκριση εκπομπών, για την οποία τελικός υπεύθυνο είναι η ΚΑΜΠΑ. Ναι, το RDV έδωσε την ε, τελική έγκριση τύπου. Το ΚΑΜΠΑ έδωσε την έγκριση τύπου για τις εκπομπές. Σύμφωνα με την κοινωνική νομοθεσία, τελικά το RDV δεν είναι αυτό που θα πρέπει να καταθέσει επίσημο αίτημα στις αρχ... γερμανικές αρχές προκειμένου να λάβουν τα σχετικά μέτρα. Όχι. Αντίστροφα. Πρώτα θα πρέπει να αποδεχτεί ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι δεν στέκει, ότι κάτι πάει στραβά σε ό,τι αφορά τη Γερμανία και το ΚΑΜΠΕΑ, το οποίο θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να μας ενημερώσει ότι αυτό θα είχε συνέπειες για την έγκριση τύπου. Δεν γίνεται ανάποδα αυτό, δεν γίνεται αντίστροφα. Εμείς ως RDV δεν έχουμε διαπιστώσει το οτιδήποτε. Η έρευνα του ΚΑΜΠΕΑ είναι αυτή που έχει να κάνει με την Opel. Ναι, αλλά γνωρίζετε τις έρευνες του Πανεπιστήμιου της Βέρνης. Και το θέμα που κρατέθηκε στο φλαμαντικό ΒΕΡΤΕ, ότι κάτι δεν πάει καλά με το Opel Safira. Αυτό μου φαίνεται σαφές. Άρα, ως ε, ο τελικός υπεύθυνο, φαντάζομαι ότι θα θέλετε να διελευκάνετε το θέμα αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι σε κάποιο βαθμό αισθάνεστε και εσείς ότι εξαπατηθήκατε ζητήσατε από τη γερμανική KBA να ολοκληρώσει γρήγορα την έρευνα αυτή και να σας ε, χορηγήσει τα πορίσματα. Κοιτάξτε εδώ κατά πόσον κάτι δεν στέκει. Αυτό θα καθοριστεί από τα πορίσματα της KBA. για το Όπελ. Εμείς ε, δεν μπορούμε βάσει ενός άρθρου να υπενηχθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, αλλά έχετε επαφές με το ΚΑΜΠΕΑ, μας λέτε. Συμμετέχετε κι εσείς στις εργασίες τους. Ξέρετε προς τα που οδεύει η έρευνα και πότε θα ολοκληρωθεί. Πότε θα ολοκληρωθεί, αλήθεια. Δεν έχουμε ακόμα οριστική απάντηση του ΚΑΜΠΕΑ για να αναλάβουμε δράση. Ναι, αλλά συμμετέχετε στις έρευνες. Ξέρετε πώς πάνε οι έρευνες. Περιμένουμε την απάντηση του ΚΑΜΠΕΑ. Δεν μπορούμε να δράσουμε, να ενεργήσουμε, ιδάλλως. Μάλιστα κάπως παθητικούς σας ε, βλέπω. Ως αρχή φαντάζομαι ότι τελικά είστε υπεύθυνοι για την ε, γενικότερη έγκριση τύπου. Φαντάζομαι ότι έχετε και κάποια αίσθηση και κάποιο αίσθημα ευθύνη ε, για την τελική έγκριση. Γιατί στη τελική ανάλυση μία είναι η αρχή η οποία μπορεί να ανακαλέσει αυτή την έγκριση τύπου. Και αυτή είστε εσείς με τη συνεργασία της ΚΑΜΠΕΑ. Δεν λέω πρέπει να σας πω ότι μάλλον κάπως παθητική κρίνω την στάση σας. Γιατί αυτό έχει προβληθεί και στον τύπο και παντού. Και το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί στους δρόμους, το έχει πολλοί κόσμος, δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται μια παραπάνω ταχύτητα αντίδρασης. Και το Opel Safira αποτελεί τμήμα της δικής σας έρευνας. Επίσης, για να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όχι, δεν αποτελεί τμήμα των δικών μα. ερευνών, το Πολυσαφήρα. Για το ερώτημα τώρα του κατά πόσον εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να ενεργήσουν. Όχι, δεν νομίζω. Εδώ η ευθύνη είναι πραγματικά για αυτόν που έδωσε την έγκριση τύπου για τι εκπομπέ. Αυτοί ξέρουν τι ακριβώς έγινε. Κατά πόσον πρόκειται για παράνομο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται κτλ. Όσο δεν έχει διαπιστωθεί τέτοια παράνομη χρήση λογισμικού, Επίσημώ δεν ναι, μπορούν να ληφθούν επίσημα μέτρα. Ανέφερα ότι η αξιολόγηση και η εκτίμηση του τι είναι παράνομη συσκευή διάταξη αναστολής είναι ένα θέμα το οποίο αποφασίζεται σε συντονισμό και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι υπόλοιπε Ευρωπαϊκέ Αρχέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκτεθειντήριε γραμμέ και αυτό στην τελική ανάλυση θα πρέπει να εναρμονιστεί στην Ευρώπη. Να είναι ενιαίοι οι κανόνες του παιχνιδιού και να μην εξαρτάται αυτό από τον καθένα, από κάθε ξεχωριστή αρχή και να μην ε, εντοπίζεται σε μία αρχή. Στη δεν είναι σαφή τα πράγματα. Ο κ. Τουγιόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την RTV που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Αν ρωτιόμουν ένα όπελ που ζητά έγκριση τύπου από την RDV. Ε, γιατί επιλέγει την RDV. Ε, αυτή την ερώτηση όμως θα πρέπει να την κάνετε στην όπελ. Όχι, εγώ εσάς ρωτάω, γιατί έχετε και ένα κάποιο marketing, φαντάζομαι κάποια στρατηγική, για να συγκεντρώνετε ακριβώς τέτοιου είδους εντολές και αιτήματα. Γιατί διευκρινίστε λίγο την ερώτησή σας. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ρωτάτε. Πώς ρυθμίζεται η χρηματοδότηση του RDW και για την έγκριση τύπου και για την ενέργεια των σχετικών ελέγχων. Η χρηματοδότηση ρυθμίζεται όπως είναι η χρηματοδότηση όλων των αρχών. Πιστοποίησης. Για κάθε υπηρεσία προβλέπεται μια τιμή η οποία θα πρέπει να καλύπτει το κόστος. Αυτό γίνεται και στην RDW. Άρα ουσιαστικά δεν έχετε οικονομικό συμφέρον αν κάποια στιγμή δεν ζητάει κανένας κατασκευαστής αυτοκινήτων έγκριση τύπου από την RDW. Όχι, επί της αρχής όχι δεν είναι σκοπός μας. Δεν εντρεθήκαμε για να προσελκύουμε εγκρίσεις και αιτήματα εγκρίσεις τύπου. Είναι το λειτουργήμά μας κοινωνικό. Και δεν είμαστε μόνο υπεύθυνοι για έγκριση τύπου. Αυτό είναι μόνο το τμήμα των ε, εργασιών μας. Θέλουμε να δραματίσουμε και ρόλο, όπως είπα στην αρχή εισαγωγικά, στην γενικότερη ανάπτυξη και νομοθεσία για τα οχήματα. Ναι, αλλά δεν ρώτησε αυτό. Δεν ρώτησε αυτό. Ένα τέταρτο των εισοδημάτων σας προέρχεται από εργαστηριακές, από τους ελέγχους εργαστηρίων που έχετε κι εσείς. Είστε από τις λίγες τέτοιες αρχές στην Ευρώπη που έχουν τέτοια εργαστήρια. Άρα από εμπορική άποψη δεν είναι ενδιαφέρον να έχετε πιο πολλού πελάτε. Αυτό θα πρέπει να το θέσω ω ερώτημα στον ε, προϊστάμενο στον επικεφαλής του RDV. Όχι σε μένα ως υπεύθυνο για θέματα εκπομπών. Η επιτέλεση και η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι τμήμα της εργασίας του RDW. Έχουμε εμπειρογνώμονες και τα εκτελούμε τα καθήκοντα αυτά με ανεξάρτητο τρόπο. Αυτό τι σημαίνει ότι όλα αυτά τα άτομα που ασχολούμαι ως ε, RDW είναι χρήσιμα για να έχουμε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίηση. Και κοιτάξτε όμω, μιλάμε πλέον με μία από τις λίγες ε, αρχές ε, πιστοποίηση που κάνει και η ίδια ελέγχου στα εργαστηριά τη. Και όταν μιλάμε για δύσκολα θέματα, όπω είναι η διατάξη αναστολή κτλ., ουσιαστικά δεν βγάζουμε παραπάνω άκρη από ότι και με του υπόλοιπου. Εξαρτάστε από την ΚΑΜΠΑ και το καθεξή. είναι την εντύπωση ότι οι εγκαταστάσει ελέγχου δεν έχουν και οποιαδήποτε θετική επίδραση σε ό,τι αφορά τους ελέγχους σε σχέση με τα όσα προβλέπει και η νομοθεσία. Αυτό είναι δήλωση ουσιαστικά. Δεν καταλαβαίνω τι ερώτηση κρύβεται σε αυτά που είπατε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας, ουσιαστικά το 2000, από το 2010 και μετά ασχολούμαστε με την ανάπτυξη της νομοθεσίας LDE. Και αυτό το κάνουμε και με την τεχνογνωσία της LDW σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται και στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Όλη αυτή η τεχνογνωσία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της νομοθεσίας, θεωρώ. Τελευταία απόπειρα, λέει ο κ. Ιούγκ. Από το τι εννοώ. Ε, λάβατε ενδείξεις ε, για διατάξεις αναστολής μας. Λέτε ότι δεν έχουμε εμπορικό συμφέρον και ότι κάνουμε λειτουργήμα. Και κανείς όλη αυτή την περίοδο δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια, κάποιος ε, έλεγχος. Κοιτάξτε, εγώ συνεργάζομαι στενά με, το, με την TNO εδώ και πολλά χρόνια. Όλα τα χρόνια που κάνω αυτό το διεθνές έργο και ασχολούμαι με τη βελτίωση της νομοθεσίας και οι εκθέσεις του TNO μου είναι γνωστές ασφαλώς και τις έχουμε κοινοποιήσει και στην Ολλανδική Βουλή ποτέ δεν έχει ανακύψει ερώτηση για επικέντρωση, για παράδειγμα, στις διατάξεις αναστολής. Και αυτό σε ό,τι αφορά και την σύσταση ελέγχων RDE, οι οποίοι υποτίθεται ότι καλύπτουν όλο το πακέτο. Σε αυτό επικεντρωθήκαμε. Ο κύριος Έγκαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρέιντερς για τις απαντήσεις του και θα ήθελα να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Ποιος είναι τελικά υπεύθυνο για να συμμορφούνται τα οχήματα με το 5.1 και 5.2 του σχετικού κανονισμού για την κανονική χρήση και για τις διατάξεις αναστολής. Ξέρω ότι εσείς τα γνωρίζετε αυτά, αλλά το διευκρινίζω για τους υπόλοιπους που ακούν ναι, μάλιστα. Ένα άρθρο ξεχνάτε, το 5-3. Ναι, αλλά εγώ ρωτάω ποιο είναι υπεύθυνο για το 5-1 και το 5-2. Στον 7-15 του 2007 ορίζονται οι βασικές προδιαγραφές. Μεταξύ άλλων ότι το όχημα θα πρέπει να πληρεί και να συμμορφούνται με τις ε, προδιαγραμμένες εκπομπές ε, για την κανονική κρίση. Ναι, το ξέρω. Ποιο είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι τα οχήματα πραγματικά συμμορφούνται. Ή αρχές που δίνουν την έγκριση τύπου βάση του κανονισμού, του θερμοστικού κανονισμού, είναι υπεύθυνε για το ότι το όχημα πληρεί τα κριτήρια. Η RDW δηλαδή. Αν η RDW κάνει τους ελέγχους στα πλαίσια του εφαρμοστικού κανονισμού του 612 του 2007 αν υπάρχει συμμόρφωση με τους ελέγχους που προβλέπονται και ποιος ελέγχει, πώς ελέγχεται ότι πραγματικά συμμορφούνται τα οχήματα. Αυτοί είναι οι έλεγχοι που εκτελούνται στους οποίους ε, παρευρίσκονται και οι τεχνικέ υπηρεσίε, δεν είναι οι τεχνικέ υπηρεσίε αυτέ που κάνουν του ελέγχου, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο ο τη εξαγωγή των ελέγχων. Αλλά σίγουρα γίνονται πάρα πολλοί ελεγχοί, πολύ πιο πολλοί από το τεστ αν RDC. Υπάρχει και, για παράδειγμα, υπάρχει και τεστ TNO. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο τεστ. Ένα τεστ περιγράφεται ως αντιπροσωπευτικό των γενικών διατάξεων για τις διατάξεις που θα πρέπει να πληρούν τα όχημα. Πιστεύω ότι τα οχήματα που εκπέμπουν εξαπλάσεις, αυταπλάσει ε, τιμές ε, εκπομπών ε, είναι, συμμορφούνται με τις Τα οχήματα τα οποία ελέγχονται τώρα, όχι το 2007 στο ΙΡΣΕ κτλ. Τότε δεν υπήρχαν προδιαγραφές για το RTE. Ναι, όχι τώρα λέω κατά πόσον ε, συμμορφούνται με τις διατάξεις για την κανονική χρήση. Εσείς ως αρχή λοιπόν που εγκρίνετε οχήματα, ήθελα να μου πείτε κατά πόσο συμμορφούνται τα οχήματα αυτά με το 51 της νομοθεσίας. Όπως σας είπα, πρόκειται για γενικές διατάξεις. Το όχημα είναι ασφαλές. Αλλά σε τι κριτήρια βασιζόμαστε. Ερωτώ λοιπόν, σε ποια κριτήρια βασίζεστε εσείς. Εμείς βασιζόμαστε στις εναρμονισμένες προδιαγραφέ που αναφέρονται στι 6-12 του 2008. Τεστ RDC. Ναι, αλλά μα αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια, ότι τα τεστ δεν πληρώνουν τις προδιαγραφέ εκπομπών και δεν συνάπτουν με το 5.1 και το μοναδικό που μπορείτε να κάνετε είναι τα τεστ lab, δηλαδή. Ναι, μόνο τα τεστ αυτά τα, τα μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το είπα ευθύ εξ αρχή. Ότι σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των προδιαγραφών γύρω 5 και γύρω 6, ναι, διακόπτω κύριο Άικαουτ. Πού λέει ότι μπορείτε να κάνετε μόνο τα τεστ NRDC. Η εκτέλεση, μάλλον ο εκτελεστικός κανονισμός αναφέρεται στην 62 του 2008 αν πληρούνται όλοι οι όροι, χορηγείται έγκριση τύπου. Άρα δηλαδή, αν βγει ένα αυτοκίνητο στον τρόπο, μετά οτιδήποτε συμβεί, συνέβη. Όχι. Γιατί ο έλεγχο ένα οχήματο, ενό πρωτοτύπου, είναι μόνο ένα τμήμα. Πέρα από αυτά υπάρχουν και κριτήρια για την παραγωγή, το COP και για το in-service conformity, σχετικές και αυτές οι προδιαγραφές επιβάλλονται λοιπόν στον κατασκευαστή προκειμένου να φροντίσει ότι το όχημα το οποίο είναι στη φάση παραγωγής ε, τα πληρεί αυτά. Ναι, αυτό το κάνει ο κατασκευαστή, αλλά εσεί πώ το ελέγχετε αυτό, για παράδειγμα για το Opel Safira, τι γίνεται. Το Opel Safira, όπω σα είπα, δεν ε, αφορά έγκριση που χορηγήσε το RDV. Ναι, αλλά εσεί είσαστε υπεύθυνοι για την έγκριση του τύπου, γιατί λαμβάνετε όλα τα τμήματα από όλε τι αρμόδιε αρχέ. Το RTV λοιπόν είναι υπεύθυνο για την τελική έγκριση του Opel Σαφύρα. Εσεί φέρετε λοιπόν την ευθύνη προκειμένου ότι ε, πλήρει όλε τι προδιαγραφέ και ότι όλοι έκαναν τη δουλειά του σωστά. Το ελέγξατε αυτό ο έλεγχος του COP και του In-Service Conformity γίνεται σε ό,τι αφορά τις εκπομπές από το ΚΜΠΑ. Γιατί η ΚΜΠΑ είναι υπεύθυνη και συνοψίζοντας τελικά, δηλαδή ο καθένας κρύβεται ε, πίσω από το δάχτυλό του. Η κυρία Εύη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω τελικά. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω Ήδη από το 2011 είχε ξεκινήσει η συζήτηση για την εισαγωγή των τεστ RDE και ήδη στον κανονισμό 715 του 2007 δηλαδή 8 χρόνια πριν οι κατασκευαστές γνώριζαν τα όρια που θα έπρεπε να σεβαστούν από το 2014 και στο εξής για το Euro 6. Εσείς πιστεύετε πως είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερος χρόνος στις κατασκευαστικές εταιρείες σας, στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ώστε να εγγυηθούμε ότι τα αυτοκίνητα θα σέβονται τα όρια και στο δρόμο, όπως ε, θα ισχύουν με τον περιορισμό του παράγοντα συμμόρφωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. τα οχήματα τα οποία ελέγχονται βάσει του Euro 6 πρέπει να πληρούν τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο Euro 6. Και προς το παρόν αυτό περιλαμβάνει μόνο τα τεστ NEDC. Αν λοιπόν τα οχήματα αυτά πληρούν τους όρους αυτούς, στην έγκριση τύπου ελέγχεται και η συμμόρφωση παραγωγής και in-service conformity. Αυτό είναι το φάσμα το οποίο ρυθμίζεται από τον νόμο στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση η εισαγωγή του RDE, που μιλάμε για το πρώτο και δεύτερο πακέτο, είναι σε λειτουργία στην παρούσα φάση, αλλά τα κριτήρια, ο παράγοντας, ε, ο συντελεστής ε, συμμόρφωσης 1,2 δεν ε, ισχύει ακόμα. Και αυτό είναι κρίμα. Είναι κρίμα που δεν ισχύει το συντελεστή συμμόρφωση ήδη σε ό,τι αφορά το γύρο 6, αλλά πολύ απλά έτσι έχει κατάσταση. Okay, grazie. Πάσα un'altra domanda. Σα ευχαριστώ. Έχω άλλη ερώτηση. Δεν έλαβα την απάντηση που περίμενα. Υπό το φως ε, της εμπειρία σα. πιστεύετε ότι στο μέλλον Οι δοκιμές RDE, δηλαδή η τεχνολογία PEMS, θα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να προσαρμοστεί ή να χειραγωγηθεί από τους κατασκευαστές για τις προηγούμενες ακροάσεις αυτό το σενάριο δεν φάνηκε να είναι τόσο μακρό, τόσο απίθανο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σα είναι δυνατόν οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων να μπορούν να χειραγωγήσουν το δοκιμέ όχι μόνο στα εργαστήρια όπως ίσως έχει να ζήτη συμβεί, αλλά και με το νέο μέσο RDE. Ως ε, κάτω σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του RDE, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Και μία από τις πτυχές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο είναι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από το SCU των οχημάτων σε ό,τι αφορά την ε, χορήγηση πληροφοριών. Δηλαδή, εμείς επιμέναμε ότι δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητη η χορήγηση των δεδομένων για τη διαδρομή για να μην λαμβάνετε και το όχημα ότι ε, πότε πρόκειται για έλεγχο αντί ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία τα ζητήσαν ιδιαίτερα οι κατοχώρες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του RDE. Και φυσικά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% ασφάλεια, αλλά τα κριτήρια τα οποία ισχύουν τώρα για το RDE θεωρούμε ότι δίνουν μια πολύ καλή προστασία και αποτρέπουν προσπάθειες και απόπειρες χειραγώγησης. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Μια τελευταία ερώτηση, σύντομα. Πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο να προβλέψουμε οι αρχές έγκρισης τύπου να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν ε, τις ε, εντός των ε, κατασκευαστικών εταιριών εγκαταστάσεις αντί για τις εξωτερικές ε, τεχνικές υπηρεσίες για το RD. Δεν ξέρω αν καλά κατάλαβα την ερώτησή σας, αλλά... Το τεστ ε, RDE είναι τμήμα του τεστ έγκρισης τύπου. Και σας είχα αναφέρει και εισαγωγικά ότι το τέταρτο πακέτο περιλαμβάνει και διεξαγωγή ελέγχων RDE και από ανεξάρτητους φορείς για χορήγηση δεδομένων για το κατά πόσον το όχημα πληρεί τους όρους. Υπάρχει λοιπόν ένας τεστ Και αν η συνθήκη, για παράδειγμα, θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου, ε, πολύ απλά τα αποτελέσματα αφορούν τις 25 βαθμούς Κελσίου, όχι τους 2 βαθμούς Κελσίου. Άρα και στο τεστ RD περιλαμβάνονται σημαντικά στοιχεία τα οποία θα ελέγχονται σε άλλους, ε, από άλλους, υπό άλλους όρους το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια του RD σε όλες τις συνθήκες. Και αυτό είναι ένα από τα ισχυρά σημεία του RD. Μάλιστα, δεύτερος ε, γύρος ερωτήσεων, ο κ. Σούλτς. Ευχαριστώ, Πέτρε Και θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά, μιας και δεν μιλάω ολλανδικά. Κύριε Ρέιντερ, σας ευχαριστούμε πολύ κατέ από τις 100 χώρες στο Βέλγιο σήμερα για να σα θέσει ερωτήματα. Ένα γερμανο. Μία ερώτηση έχω να σας κάνω. Την οποία την έθεσα και χθε στους συναδέλφου σα και σήμερα το πρωί. Μία τεχνική ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την προστασία των εξαρτημάτων. Μία ερώτηση να επαναλάβω και θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς κατά πόσον πιστεύετε ότι οι τάξεις αναστολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προστατεύονται εξαρτήματα όπως έμεσα ή άμεσα προβλέπεται στην νομοθεσία. Αυτό γενικώ πώς, πέρα από αυτά που γνωρίζουμε για το πώς μπορεί να εκμεταλλεύονται στην τάξη αναστολή οι κατασκευαστές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. οι κατασκευαστέ φέρουν την ευθύνη του ασφαλώ. και θα πρέπει να φροντίζουν οι συσκευέ που χρησιμοποιούνται για να περιορίζονται οι εκπομπέ λειτουργούν σωστά. Αν και κάποιο λόγο, κάποιο εξάρτημα του συστήματο αυτού του περιορισμού των εκπομπών ε, τίθεται εκτό λειτουργία γιατί προκύπτει μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να προστατευτεί ο κινητήρας, αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται Προφανώ. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το σύνολο του συστήματο θα πρέπει να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπομπέ τελικά κατά μέσο όρο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο να παραμένουν κατά απορισμένα επίπεδα. Και στο RDE χρησιμοποιούνται κάποια εργαλεία μέσης διαμόρφωσης, διαμόρφωσης μάλλον του μέσου όρου. Δεν λέμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές δεν θα υπάρξει κάποια εχμή. Το ότι ένα σύστημα ε, απαντεργοποιείται κατά διαστήματα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβλέπεται ως δυνατότητα. Αλλά δεν είναι δυνατό το συνολικό σύστημα για κάποιον ανεξήγητο λόγο να τύφεται εκτός α, λειτουργίας για την εξοικονόμηση, για παράδειγμα, μόνο καυσίμου. Αν ερμηνεύσω λοιπόν αυτά που μας είπατε, αυτά που τους τελευταίους μήνες μαθαίνουμε για το πώς οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν την προστασία των εξαρτημάτων για κάποιες θερμοκρασίες, για πενταργοποίηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. διάστημα. Αυτά τα θεωρείτε λοιπόν. Λανθασμένη χρήση των όσων αποσκοπεί η προστασία των εκκρατημάτων αυτών. Καλά κατάλαβα. η αξιολόγηση, η εκτίμηση του κατά πόσον η επενεργοποίηση κάποιου τμήματος ε, του συστήματος περιορισμού των καυσαρίων επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες και γι' αυτό είναι πολύ περίπλοκο να κρυθεί και να αξιολογηθεί. Δεν μπορώ στον αέρα να κρίνω. Μια σωστή λοιπόν έρευνα θα χρειαζόταν για τους λόγους, τις αιτίε διαμόρφωσης της στρατηγικής και της προσέγγισης αυτής και κατά πόσο είναι αποδεκτή ή όχι. Αυτό θα προϋπέθεται και την απαραίτητη τεχνογνωσία και την δυνατότητα να τεθούν πολλά ερωτήματα προς τον κατασκευαστή. Γιατί γίνεται αυτή η επενεργοποίηση, δεν είναι απλή απάντηση. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε έτσι κατά πόσον αυτό επιτρέπεται ή όχι. Όχι. Θα πρέπει να ξέρουμε και τα επιχειρήματα και να γνωρίζουμε σε βάθος την τεχνολογία. Και κατά πόσον πρόκειται για μία διάταξη η οποία είναι παραδεκτή ή όχι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Μία άλλη ερώτηση προς μία άλλη κατεύθυνση, επιτρέψτε μου στο τελευταίο λεπτό. Κάνετε και ενός είδους εποπτεία της αγοράς για τα οχήματα που έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου και δειγματοληπτικά περνούν από ελέγχους. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν πόσους τέτοιους ελέγχους έχετε κάνει δειγματοληπτικούς και στους ελέγχους αυτούς που έχετε κάνει τους δειγματοληπτικούς μάλλον έχουν αυξηθεί αυτοί οι έλεγχοι αριθμητικά μετά από το σκάνδαλο του τελευταίου έτους. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να διακρινούμε μεταξύ δύο είδων εποπτεία αγοράς. Όταν μιλάμε για παρακολούθηση της αρχής που χορήγησε την έγκριση τύπου του κατασκευαστή, η αρχή αυτή έχει καθήκον να ερευνά κατά πόσον η συμμόρφωση της παραγωγής γίνεται με σωστό τρόπο τα πλαίσια της κατασκευής και παρακολουθεί ότι γίνεται η παραγωγή αυτή, η κατασκευή αυτή βάσει των κανόνων. Ιδάλλως θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Πέραν αυτού, εξετάζεται κατά πόσο τα οχήματα τα οποία ήδη είναι σε χρήση και έχουν ξεπεράσει τα 160.000 χιλιόμετρα για παράδειγμα, πληρούν ακόμα τα κατήρια αυτά. Αυτό είναι τμήμα της έγκρισης τύπου. Όταν μιλάτε λοιπόν για παρακολούθηση της αγοράς, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Το RDW δεν το κάνει αυτό. Δεν παρακολουθεί την αγορά. Δεν ελέγχουμε τα οχήματα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην Ολλανδική αγορά. Αν μιλάτε τώρα για τον έλεγχο που γίνεται στο πλαίσιο του TNO, που κάνει κάποιον έλεγχο για να διαπιστώσει την ε, επίδοση των ε, χημάτων σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν βενζίνη και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν δίζελ. Για παράδειγμα, τι εκπομπές έχουν σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Η πρόεδρος. Ποια αρχή όμως, ποια υπηρεσία τελικά κάνει την υποπτήρια της αγοράς στην Ολλανδία. Το Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος η επιθεώρηση μεταφοράς μεταφορών κάνουν τεστ στον δρόμο. Αυτό θα έπρεπε να το θέσετε ως ερώτημα προς το Υπουργείο. Θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παλούτσι. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις απλές και σύντομες. Έτσι θα κερδίσουμε το χαμένο καιρό. Χτες η αρχή έγκριση τύπου της Ιταλίας αναφέρθηκε σε υποθέσεις όπου μη εγκεκριμένα αυτοκίνητα στην ουσία, στη συνέχεια μάλλον έλαβαν έγκριση τύπου από άλλες εθνικές αρχές. Γνωρίζετε και εσείς αντίστοιχες περιπτώσεις. Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στην Ολλανδία. Δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή γιατί πολλοί απλά δεν το ξέρουν να σας απαντήσω αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ για τη μία απάντηση. Και η δεύτερη είναι περισσότερο είναι μου και όχι ερώτηση. Η δική σας αρχή είναι η τρίτη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα μοντέλα που, δίνονται, που δίνει, χορηγεί την έγκριση τύπου, αν και στην Ολλανδία δεν υπάρχει ε, κατασκευαστική εταιρεία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η φοβερή σας επιτυχία. Νομίζω ότι η W είναι αξιόπιστος εταίρος και επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της. Και νομίζω ότι βάση της ποιότητας, της τεχνογνωσίας και της αποτελεσματικότητας αποτελεί μια επιτυχία. Σας είπα ότι δεν κάνουμε οποιαδήποτε εμπορική προώθηση ή τέτοιες ε, έγκρισης τύπου. Θεωρούμε ότι είμαστε μια οργάνωση τέτοια οποία με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο μπορεί να κάνει τους ελέγχους, να χορηγεί εγκρίσεις τύπου. Ενδεχομένω αυτό να οδηγεί τους κατασκευαστές στην υποβολή αιτήματο στην RDW στην Ολλανδία για την ενέργεια των ελέγχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Αγιάλα Σέντερ κατεύθυνση. Με εκπλήση που το 2015 η Τέσλα που μόλις είχε εμφανιστεί, είχε πέσει από τον ουρανό, ε, ε είχε ε, οχήματα και δεν ξέρω αν τα είχατε εσείς ε, εξετάσει καθόλου. Μετά για την έκθεση την οποία θα υποβάλατε, θα θέλω να σας ρωτήσω πώς μοιραστήκατε τη δουλειά σας εσείς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών. Ποιος πλήρωσε τι, πώς συνεργαστήκατε ε, ένα κρατικό ερευνητικό κέντρο που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προπολισμό ε, και ε, εσείς. Πώς συνεργαστήκατε, πώς επιμερίσατε το έργο. Ε, σε αυτή την ε, εργασία που κάνετε, για την έκθεση που θα υποβάλλετε. Ε, Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω επαρκώς στην ερώτησή σα γιατί είναι πάντα δύσκολο να καταλαβαίνω Ακριβώ τι με ρωτάτε. Ναι, σε ό,τι αφορά την Τέσλα. Την Τέσλα Πρόκειται για ένα κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήσαμε έγκριση τύπου για πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Εδώ δεν υπάρχουν εκπομπές, άρα έτσι είναι λίγο πιο απλή η κατάσταση. Πρόκειται για μία έγκριση τύπου την οποία χορηγήσαμε προς την Τέσλα. Δεν ξέρω, ρωτήσατε και κάτι άλλο. Ναι, ε, πώς συνεργαστήκατε και πώς πρόκειψε η χρηματοδότηση ε, για κάθε ένα από τους φορείς ε, που ασχολήθηκαν με την έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών και εσείς. Ε, πώς συνεργαστήκατε εσείς δύο, αυτό ρωτούσα. Ε, εν αναμονή της έκθεσης την οποία θα υποβάλλετε στο Ολλανδικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζω. Ποιος πλήρωσε τι, πώς μοιραστήκατε τα καθήκοντα κλπ. onderzoeken die, eh, die wij hebben gedaan, komen uit eigen... Οι έρευνε που κάναμε εμεί ε, χρηματοδοτούνται από του δικού μα πόρου. Όλοι οι έλεγχοι που έγιναν και όλοι οι επιμέρους έλεγχοι που χρειάζονται χρηματοδοτούνται από την RDW. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον από αυτά που μου είπε ο συνάδελφος, γιατί δεν είναι δικός μου, δεν είναι, ειδικότητά μου. Αυτή, δεν ξέρω μήπως θέλετε να πάρει το λόγο και ο συνάδελφός μου να πει κάτι παραπάνω. Είπατε ότι το κέντρο ευνών σας βοήθησε πάρα πολύ. Το είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας. Ε, με ξέπληξε πώς είναι το να σας βοηθήσει. Γι' αυτό το λόγο ρωτάω. Η JRC είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα που υποστηρίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία αντι είναι μεγάλο τμήμα που κάνει αναλύσεις μοντελοποίηση για τι φορτές συστήματα μέτρηση εκπομπών. Και όλα αυτά αξιολογούνται λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα εμείς για την βελτίωση των συστημάτων αυτών. Συνεργαζόμαστε με τον TNO, το οποίο συνεργάζεται με το Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος με τη σειρά του. Το χρησιμοποιώ με πολύ ευγνωμοσύνη για να χρησιμοποιήσω και την ε, τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνολογία που διατίθεται στον TNO για την νομοθεσία των, ε, του RDE. Ευχαριστώ, κύριο Γκίζικε, για δύο σλότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επανέλθω στα θέματα ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ερώτηση 1 λέτε ότι δεν υπήρχε ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και κάπως ενοχλούμε και αγανακτώ γιατί ο Ιταλός συνάδελφος άλλα μας είπε ότι υπάρχει τέτοια ανταλλαγή απόψεων. Εσύ μας λέτε ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Και πληροφοριών. Οι πληροφορίες των τεχνικών υπηρεσιών ουσιαστικά δεν ανταλλάσσονται αλλά οι πληροφορίες μεταξύ των υπηρεσιών έξις τύπου ανταλλάσσονται. Τη στιγμή λοιπόν που χορηγείται προς την τεχνική υπηρεσία μία έκθεση η οποία καταδεικνύει ότι ένα όχημα δεν μπορεί να λάβει έγκριση τύπου γιατί δεν πληρεί τα κριτήρια, μπορεί να ενημερωθούν οι υπόλοιπε αρχέ έγκριση τύπου. Αυτή η επικοινωνία γίνεται. Σας ευχαριστώ. σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου, πάντα τίφερε το θέμα της ε, οικονομικής ανεξαρτησίας και εδώ σε σχέση με τη ΣΥΠΑ αναφέρεται ότι η έμεση χρηματοδότηση από τους κρατικούς πόρους στην Αμερική αποτελεί το καλύτερο σύστημα. Αν συγκρίνουμε λοιπόν το αμερικανικό σύστημα με το ευρωπαϊκό σύστημα, γιατί στο ευρωπαϊκό σύστημα έχουμε άμεση εξάρτηση κατά 25% της χρηματοδότησης, δεν πιστεύετε για παράδειγμα ότι το ευρωπαϊκό σύστημα σε σχέση με το αμερικανικό στερεί κάπως. Η χορήγηση έγκρισης τύπου είναι δύσκολο... Μάλλον, κάθε σύστημα έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό σύστημα με τις προσαρμογές του όπως γίνονται τώρα στο Συμβούλιο. Είναι αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τα οχήματα. Απαιτεί συνεργασία μεταξύ των κρατών μέσω, μεταξύ των υπηρεσιών χορηγήσης έγκρισης τύπου και υπάρχουν αυτά τα συστήματα λοιπόν, αυτά τα κοινά στοιχεία. από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζονται και σαφεί προδιαγραφέ και κατευθυντήριε γραμμέ για τη συνεργασία. Και νομίζω ότι πλέον η πρόταση που βρίσκεται επιτάπητο στο Συμβούλιο και με τα peer reviews και με τους ελέγχους και με τους ελέγχους πιστοποίησης βελτιώνει το ευρωπαϊκό σύστημα. Το σύστημα των Αμερικανών της αυτοπιστοποίησης ουσιαστικά για άλλα μειονεκτήματα. Το όχημα μπορεί να έχει ήδη βγει στο δρόμο και να διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτό ασφαλώς έχει μεγάλες συνέπειες. Και αυτός είναι ένας άλλος κινδύνος για τους κατασκευαστές και για το ίδιο το σύστημα. Και οι ποινές είναι πάρα πολύ σκληρές και αυστηρές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ανισόρροπη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Πρώτα τελευταία τεχνική ερώτηση, την οποία την έθεσα και στους Γάλλους συναδέλφους σας σήμερα. Το θέμα της ακρίβειας μετρήσεων των PEMS, των φορτών συστήματων μετρήσεων εκπομπών. Ο, ο Γάλλος συναδελφός σας ε, μίλησε για 100% ακρίβεια με μία ανοχή 20% επιβεβαιώνεται αυτές τις ε, εκτιμήσεις. οι συσκευές PEMS για τις εκπομπές πέρα από τις συσκευές PEMS που είναι για τα σωματίδια συγκεκριμένα για το διοξείδιο του αζότου η ανοχή είναι περίπου 2% Υπάρχουν άλλα όρια ανοχής για τους ελέγχους και υπάρχουν και άλλα κριτήρια και συνολικά. Η συνολική αβεβαιότητα για τα οχήματα με σύστημα PEMS ορίζονται στο 0,5 συνολικά σε ό,τι αφορά την συσκευή 0,2 λοιπόν και για το συνολικό πακέτο 0,5. Και αυτά είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το JRC. Σας ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση. Πέντε δεύτερα. Ήταν εδώ και ο, υπουργός, ε, ο Γερμανός Μεταφορών εδώ. Αν είχατε μια ερώτηση να του κάνετε, ποια θα ήταν αυτή. Δεν θα είχα ξεκάθαρα κάποια κατεύθυνση να ακολουθήσω, αλλά κοιτάξτε. Φυσικά θα ήθελα μια γενικότερη συνεργασία μεταξύ των μερών. Αυτό θα ήθελα να προτείνω, αλλά όχι κάποια συγκεκριμένη ερώτηση δεν θα είχα να του κάνω. Η ε, κυρία Γκρίφιν. Uh, thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης ε, ανάμεσα στις διάφορες αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο τροφοδότησε αυτήν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οι διάφορες αρχές ερμηνεύουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία με διαφορετικό τρόπο, με πιθανές εξαιρέσεις ε, όσον αφορά την απαγόρευση συσκευών αναστολής. Ε, αναπερίπτωση, εν μέρει απαντήσατε, αλλά συγκεκριμένα στην ερώτηση 12 δέχεστε ότι το σβήσιμο του συστήματος ελέγχου εκπομπών μετά από 20 λεπτά λειτουργία στο κινητήρα απαγορεύεται και είναι απαγορευμένη συσκευή αναστολής. Ο Ιταλός συνάδελφος ωστόσο δεν, φάρισε, δεν θεώρησε τον αρκετά ύποπτο αυτό ώστε να ξεκινήσει έρευνα για το θέμα αυτό και δεν παρέτεινε τη στάνταρ διάρκεια μια της δοκιμής για να επαληθεύσει αν αυτές ε, οι καταγγελίες επιβεβαιώνονταν ή όχι. Εσείς μπορείτε αυτό να το σχολιάσετε και μπορείτε μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορετική προσέγγιση ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, τύπου. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για το κατά πόσο μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να την ε, αποφασίσουμε από κοινού και αρμονισμένα στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές, οι αρχές έγκρισης τύπου θα έχουν ε, η καθεμία την άποψή τη για το ποια κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, αλλά για μια συνολική, για παράδειγμα, απόφαση απανεργοποίησης ε, μιας ε, συσκευής μετά από 20 λεπτά δεν μπορώ να απαντήσω κατά πόσον είναι απαραίτητο αυτό για την προστασία του κινητήρα ή όχι. Αλλά, αλλά πρόκειται για μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε και θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από τον κατασκευαστή για τους λόγους που τον οδηγούν στην απενεργοποίηση αυτή και να μπούμε σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας για να δούμε κατά πόσο αυτό περιλαμβάνεται και θα μπορούσε να καλυφθεί από τις εξαιρεσει για τι διατάξει αναστολή. Φυσικά, ε, τα κράτη-μέλη και οι τεχνικέ υπηρεσίες μπορούν να έχουν η κάθε μία την άποψή τη και την τοποθέτησή τη Άρα στην Ευρώπη προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό τόπο. Και αυτά θα έπρεπε να δημορφωθούν υπό τη μορφή καταθετηρίων γραμμών προς όλες τις ε, τεχνικές υπηρεσίες και τι υπηρεσίες έγκρισης τύπου. Εναρμόνιση λοιπόν. Ευχαριστώ. Είστε σίγουρος ότι αυτά τα βήματα θα οδηγήσουν ε, στο να ε, δυσκολέψει η δυνατότητα να κλέψουν, ας πούμε, τα κρατη να προβούν σε απάτες. Αυτό ελπίζω, αυτό θέλω. Είμαστε το μέσο της διαδικασίας αυτής ακόμα. Δεν υπάρχει ακόμα σχετική ολλανδική έρευνα, αλλά σίγουρα θα συμμετέχουμε κι εμείς στη συζήτηση. Θέλουμε να καταλήξουμε σε καλές κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα υποσχέται και τέτοιες κατευθυντηρίες γραμμές. Προκειμένου από κοινού να αποφασιστεί πώ θα γίνεται η ανείχνευση των διατάξεων αναστολή. Γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων. Στην τελική ανάληψη, θα έπρεπε να είναι και νομικά δεσμευτικέ αυτέ οι κατευθυντηρίες γραμμέ. Και αυτά θα πρέπει να δοθούν ως κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρχές έγκρισης τύπου και τις τεχνικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Κύριε Χερμπράντη, θα πάρετε πάλι το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την πολιτική εμπειρία του κυρίου Ράιντερ σε ό,τι αφορά τη διαδικασία RDE Είπατε ότι στην αρχή του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν καινούργια τέσσερα και μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 χρειάστηκε. Τέσσερα χρόνια λοιπόν για να διοργανωθούν οι σχετικές ημερίδες και τελικά χρειάστηκαν άλλα πέντε χρόνια για να ετοιμαστεί το πρώτο πακέτο RDE. Τον 2010 θεωρούσαμε ότι αυτό θα έπαιρνε μόνο δύο χρόνια. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία πήρε σχεδόν 10 χρόνια. Εξηγήστε μας, γιατί τεχνικός πώς δεν είναι και τόσο περίπλοκα τα πράγματα. Να, το γιορτώσω. Τεχνικός πώς είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα αυτό. Όχι τόσο δύσκολο που να χρειάζονται 10 χρόνια. Αν σας κλείσουμε σε μία αίθουσα και σας δίνουμε και λίγο φαγητό μαζί με τους εμπειρογνώμονες, μέσα σε ένα χρόνο δεν μπορεί, να τα βγάλετε πέρα. Ναι, και εμείς αυτό είχαμε ελπίσει. Αυτό ελπίζαμε. Αυτή τη φιλοδοξία είχαμε. Το 2011 ξεκινήσαμε το RDE και το RDV το 2011. Και χρειάστηκε καιρό να προσανατολιστούν ε, προς την διακατεύθυνση οι αρχές εγκρισής τύπου, οι κατασκευαστές, οι αρχές, οι τεχνικές υπηρεσίες κτλ. Ήταν πολιτικό το θέμα. Κοιτάξτε, εκ των υστέρων με όλα όσα γνωρίζουμε είναι εύκολο να κρίνουμε, αλλά τότε η κατάσταση ήταν διαφορετική. Τότε λοιπόν λέγαμε ότι το όχημα θα πρέπει να συμμορφούνται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτό που λέμε και ξαναλέμε τώρα. Και αυτό το ελέγχαμε με μια εναρμονισμένη μέθοδο, με το RDC. Αυτό υποτίθεται ότι αποτελούσε αναπαράσταση είναι στο Q-test. Και τα αγόρια λοιπόν αυτά βασιζόντουσαν στους ελέγχους αυτούς. Τότε όμως εκφράστηκε η εξή σκέψη. Τα όρια αυτά είναι ανεξάρτητα από τον τεστ. Θα μπορούσε να γίνει και άλλο τεστ. Και αυτό ήταν λοιπόν μια αλλαγή τη νοοτροπία και γι' αυτό καταφέραμε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη του RDE. Ναι, αλλά μιλάμε για τον Ιανουάριο του 2011. Πέντε χρόνια λοιπόν χρειάστηκαν από τότε που διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζονται καινούργια τεστ. Πέντε χρόνια δεν έγινε τίποτα. Ξαναρωτώ λοιπόν. και οι κατασκευαστέ δηλαδή τελικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο γιατί αναφέρατε ότι και αυτοί συμμετείχαν. Πείτε μας όμως. Υπήρξαν και άλλα συμφέροντα πέρα από τα τεχνικά συμφέροντα. Έγιναν πολιτικά παιχνίδια από τα κράτη-μέλη, από τους κατασκευαστές και ούτω καθεξής για να διαρκέσει επαόριστον αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση είναι δύσκολο να απαντηθεί. Εγώ παρακολούθησα την διαδικασία αυτή εξ αρχής. Και συμμετείχα ενεργά για να γίνουν βελτιώσεις στη διαδικασία αυτή. Αλλά η ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης χρειάστηκε δύο τρία χρόνια ουσιαστικά. Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μοντέλο για το πώς ε, μπορούν να αναλυθούν τα δεδομένα με ένα PEMS και να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο όριο. 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο σε ό,τι αφορά την εκπομπή διοξιδίου του αζότου. Αυτό λοιπόν είναι εργαλείο τυποποίηση. Πιο σωστό από το εργαλείο αξιολόγηση και είχαμε διάφορε εναλλακτικέ, ε, όπω για παράδειγμα τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας για τα βαρέα χρήση ε, φορτηγά. Αλλά σε ό,τι αφορά τα γραμμάρια ένα χιλιόμετρο, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μουνιφά. Ε, Στα γαλλικά θα μιλήσω. Εγώ θέλω να συνεχίσω από το όσα είπε η συνάδελφος Γκρίφιν και για το γεγονός ότι είναι δύσκολο να εναρμονιστούν οι διάφορες ε, εθνικές αρχές όσον αφορά τα θέματα συντονισμού ε, για το τι είναι και τι δεν είναι μια συσκευή αναστολής. Η έκθεση που το υποβάλλεται στις αρχές σας θα γίνουν επί τη βάση των κατευθυντηρίων γραμμών Ε, για τις συσκευές αναστολής. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει μια ενημέρωση για το τι είναι και τι δεν είναι αυτές οι συσκευές Και έπειτα, για να φτάσουμε σε αυτή τη φάση, δεν θα ήταν ο καλύτερο τρόπο να περάσουμε από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που θα ήταν υπεράνω των εθνικών οργανισμών και θα, που θα μπορούσε να εναρμονίσει, να ρυθμίσει και να αποφασίσει σε περίπτωση που χρειαστεί διατησία, ας πούμε, για την, ε, το, τι, τους ορισμούς ή οτιδήποτε. Για την πρώτη σας ερώτηση. Ναι, η εμπειρία από διάφορα προγράμματα και από το πρόγραμμα ελέγχου το οποίο εφαρμόσαμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτυχθούν καλές κατευθυντήριες γραμμές για, τα, για τις διδάξεις αναστολής. Αν, λοιπόν, ως αποτέλεσμα αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα σύγκρισης τύπου, αυτό θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το Euro 5, για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι καταπίπτουν οι προδιαγραφές αυτές και ότι δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα γύρω 5, θα ακολουθεί το Euro 6 ως πρότυπο και θα προσαρμοστούν τα οχήματα γύρω 5. Και νομίζω ότι κυρίω στο αυτό το τελευταίο θα πρέπει να εστιαστούμε και να επικεντρωθούμε. Τώρα, κατά κατά πόσο θα να αναλυφθεί η δράση, σίγουρα θα πρέπει να είναι κοινή αυτή η δράση. Δεν είναι δυνατόν να αναλάβει δράση μία μόνο αρχή κατά ενός μόνο κατασκευαστή. Όχι, θα πρέπει να είναι κοινά κριτήρια για το τι είναι υπεύθυνο, τι δεν είναι υπεύθυνο, τι αποτελεί προστασία του κινητήρα και τι όχι. Για το δεύτερο ερώτημα. κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει κάποιος επόπτη σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου. Νομίζω ότι στην παρούσα πάση το Συμβούλιο συζητιέται ο νέος κανονισμός για την έγκριση τύπου και για την εποπτεία της αγοράς. Οι συζητήσεις αυτές είναι σε εξέλιξη. Μιλούσα για ανεξάρτητη αρχή. Αυτό προτείνεται από την Κομισιόν, δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Εγώ ε, μιλούσα για μια αρχή του τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Σιδηροδρόμων, για παράδειγμα. Αν επανέλθω στην νομοθεσία για τις εκπομπές, στο τέταρτο πακέτο του RDE περιλαμβάνεται ε, μια περιγραφή των ανεξάρτητων μερών. Άρα, υπάρχει ένα στοιχείο εποπτείας της αγοράς ε, στην έγκριση τύπου. Νομίζω ότι αναφέρεται στην ερώτηση για την νομοθεσία που βρίσκεται στο Κοινοβούλιο για την έκρηση τύπου και ότι κάποιοι στο Κοινοβούλιο θα ήθελαν να δημιουργηθεί ε, μια ανεξάρτητη αρχή για την παρακολουθή της αργοράς στην Ευρώπη. Κατά πόσον είσαστε υπέρμαχος της ιδέας αυτής. Είπα ευθύ εξ αρχή ότι δεν είμαι ειδικό για τι διαπραγματεύσει που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο. Άρα πρέπει να γενικολογήσω και να είμαι πολύ προσεκτικό. Είμαστε υπέρ πάντω όλων των βελτιώσεων που έχει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα διοργανωθεί και ένα είδο επιτροπή, ανεξάρτητης που θα ε, έχει διαιτητικό ρόλο για τις δραστηριότητες των αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών αρχών. Είμαστε υπέρ λοιπόν αυτής της προτάσεις. Μάλιστα. Ο κύριος Φαϊκάουτ, τελευταίος. Σας ευχαριστώ. Για να συνοψίσω θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, διεξαγάγεται η όλη διαδικασία για να καταλήξουμε σε έναν ορισμό για τη διατάξη αναστολή. Για παράδειγμα, η Ιταλία για τη Fiat λένε ότι για παράδειγμα δεν υπάρχουν διατάξει αναστολή. Πώς ε, γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων, Πώ γίνεται η συζήτηση αυτή πολύ απλά στην παρούσα φάση. Η συζήτηση θα λάβει χώρα σε μια ξεχωριστή ομάδα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής με υποδομάδα της ομάδας αυτής που ασχολείται με την παρακολούθηση της αγοράς. Ναι, όχι, θέλω να μου πείτε για την να αναστολή, συγκεκριμένα. Αν οι Ιταλοί και ο κύριος Χουπέσερ μπέρδευε τον εαυτό του με τη Fiat, καταλαβαίνετε. Αν οι Ιταλικές αρχές δεν δίνουν δεδομένα, απλά αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία μας δεν υπάρχουν μεταξύ στολής και είμαστε στην ομάδα εργασίας. Τι θα γίνει. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναφέρει στις κατευθυντήριες γραμμές ότι αυτά είναι τα κριτήρια και θα πρέπει να τηρήσει και η Ιταλία. Οι Ιταλοί χθε είπαν ότι εντάξει δεν ε, απενεργοποιούνται οι συσκευέ αυτέ, ε, πάνε στο 70% και ότι αυτέ δεν αποδέχονται και ουσιαστικά αποδέχονται ότι δεν πρόκειται για τέτοια τάξη αναστολή. Τι θα γίνει λοιπόν, αν οι Ιταλοί βγουν και πούν ότι δεν υπάρχουν τάξη αναστολή. Αυτό προέκυψε από την έρευνά σα. Θα το αποδεχτείτε αυτό στη συζήτηση. Στην παρούσα φάση γίνεται συζήτηση των γερμανικών αρχών με τι Ιταλικέ αρχέ και διαμεσολαβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σε ό,τι αφορά τον συντονισμό της αξιολόγησης, οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελπίζουν να καταστούν υποχρεωτικές, ελπίζεται. Εγώ θεώρησα ότι είναι δεδομένο αυτό, κοιτάξτε. Οι κατευθυντήριες γραμμές από πλευράς νομικής είναι διαφορετικές από την από την νομοθεσία. Ναι, αλλά ξέρετε ότι από το 98 χρησιμοποιούνται διατάξεις αναστολής στην Ευρώπη. Μέχρι το 2015 δεν έγινε τίποτα. Όλοι έμειναν έκπληκτοι παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν γνωστό για τα φορτηγά. Τι διαφάνεια υπάρχει, τι συμφέροντα έχουν τα κράτη-μέλη, πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε, τι θα γίνει και πότε και πότε θα έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πόρισμα θα πρέπει να περιμένουμε την κοινή διαμόρφωση κριτηρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κατευθυντήριες γραμμές. Εγώ βλέπω να συμβαίνει την πρόοδος. Ναι, αλλά πόσο θα πάρει ακόμα. Κοιτάξτε, ασκείται έντονη πίεση για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία αυτή. Αυτή την ερώτηση όμως θα πρέπει να την κάνετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβληθούν οι καθημερινές γραμμές. Ε, εγώ, η RDW, μπορεί να έχουμε μία εικόνα για το τι θα πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί όμω αυτό. Θα πρέπει από κοινού να τα διαμορφώσουμε όλα αυτά και χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα καταθέσει τα κριτήρια αυτά. Κύριε Έκχαουτ, ο Επίτροπος ε, υποσχέθηκε να τα έχει ολοκληρώσει όλα αυτά μέχρι το τέλη του έτου. Ελπίζω να ανταποκριθεί στι δεσμεύσει αυτέ και όλα τα κράτη-μέλη ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα υποβάλουν τα κρατημέλη. Εδώ πέρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με έλλειψη διαφάνειας. Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ναι, θα χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, για την απάντηση που δώσατε στα πολλαπλά ερωτήματα. Ολοκληρώσαμε μια μισή ημέρα ακροάσεων όπου μάθαμε πολλά, αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν εκκρεμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που συμμετείχατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολη η σημερινή ημέρα και ήταν δύσκολη και η εβδομάδα αυτή. Έγιναν πάρα είχαμε και πολλές ε, συνεδριάσεις επιτροπών. Ήταν πολύ επικοδομητικές αυτές οι συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ και καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Την επόμενη Δευτέρα έχουμε τη Fiat.